Συνάδελφοι, αν θέλετε καθίστε για να ξεκινήσουμε. Ένα θερμό όρισμα σε όλους σας, συνάδελφοι. Αγαπητοί συμπρόεδρε, κυρία Λούγκερ, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσκαλεσμένοι μας και ομιλητές μας. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω σήμερα στην τρίτη συνάντηση της μεικτή ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου της Europol, την οποία έχει συνδιοργανώσει το Αυστριακό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό. Βεβαίως λαμβάνει χώρα στην, στο ημικύκλιο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, συνάδελφοι, χαίρομαι που 67 εθνικοί βουλευτέ έχουν προσέλθει σήμερα εδώ και εκπροσωπείται 37 κοινοβούλια και βουλές και 27 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες, από και προς, αλλά θα πρέπει να πω ότι επειδή δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση της μειχτής ομάδας, ε, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία η ομάδα αυτή και οι συνεδριάσει τη για την επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε με τα κράτη-μέλη. Διότι αφορά τα θέματα της Europol, ε, τη Ευρωπόλ, έναν οργανισμό που μα ενδιαφέρει πολύ στο Ευρωκοινοβούλιο. Από τη δική μα τη σκοπιά και παρακολουθήσαμε την εξέλιξή της από τη γέννησή της και την ε, το πώς μεγάλωσε. Νομίζω ότι θα παραδεχτείτε κι εσείς ότι μέσα από τους μηχανισμούς λογοδοσίας που έχουμε κατασκευάσει, η σκληρή δουλειά του οργανισμού και του προσωπικού της έχει δώσει αποτελέσματα και μάλιστα επιτυχή. Η σημερινή λοιπόν συνεδρίαση εξελίσσεται σε μια καλή διαδικασία λογοδοσίας και ελέγχου και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωκοινοβούλιο. Σα καλωσορίζω και πάλι θερμά λοιπόν και ελπίζω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεδρίαση σήμερα και αύριο. Θα ήθελα να σας πω ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν διερμηνία σε όλους. Ήταν ένα πρόβλημα στην προηγούμενη συνεδρίαση αυτό και επειδή είναι εβδομάδα κοινοβουλευτικών επιτροπών αυτή, έπρεπε να δώσουμε μια προτεραιότητα στις επιτροπές και στις εργασίες τους. Είναι όμως πιστικό και το πρόγραμμά μας, ε, γιατί είναι η τελευταία χρονιά πριν τις ευρωεκλογέ για τις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου στη θητεία μας. Συνάδελφοι, λοιπόν, ανέφερα την ευρωπολο ως οργανισμό. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, που δεν είναι πλέον τόσο νέα, ίσως να αισθάνεται ότι έχει αναλάβει από καιρό καθήκοντα, για την ε, μεγάλη θέση της. Καλωσορίζω την Κάθριν Τεμπόλε, η οποία ανέλαβε 1η Μαΐου του 2018. Θα την έχετε συναντήσει πολλοί από εσά και θα ήθελα επισήμω στη σημερινή συνεδρίαση να την καλωσορίσω ξανά και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του Ευρωκοινοβουλίου για τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε ως τώρα. Σας στηρίζουμε πλήρως και εσάς και την ομάδα σας και τη δουλειά που κάνετε για την ασφάλεια. Σήμερα θα έχουμε συζήτηση για το πολιετές πρόγραμμα εργασίας 2019-2021 με την κυρία Δεμπόλ και μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Πέκνα, τον ε, πρόεδρο της ε, ομάδας διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ και του κυρίου Τσφετάνοφ, του συμπροέδρου της μεικτής ομάδας. Θα συζητήσετε αύριο θέματα για την δίωξη οικονομικού εγκλήματος, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τον κύριο Ράισενμπικ που είναι από, το από την Ολλανδική Εισαγγελία και, τα σχετική, τη σχετική υπηρεσία συντονισμού ε, καταπολέμησης οικονομικής τρομοκρατίας και την κυρία Ντεμπόλ. Επίσης ο κ. Βερκόφσκι που είναι ε, βοηθός ε, επόπτης για θέματα EDPS ε, και θα μάθετε από αυτόν τα τελευταία πορίσματα και δραστηριότητες για τα θέματα προστασίας δεδομένων. Επίσης ο Επίτροπος Κιν που είναι υπεύθυνο για την Ένωση Ασφάλειας θα σας δώσει μια ομιλία, θα εκπονήσει μια ομιλία αύριο. Θα ήθελα να σα πω ότι η Τρόικα των Προεδριών είχε οργανώσει μια προπρασκευαστική συνεδρίαση το πριν από αυτή τη συνεδρίαση. Και εκεί συζητήσαμε και την εκπροσώπηση της Δανίας στις συνεδριάσεις της ΜΟΚΕ. Η εκπροσώπηση θα γίνει αύριο το πρωί ε, βάσει της απόφασης που είχε ληφθεί τον περασμένο Μάρτιο και όλοι, έχουν, όλοι οι εκπρόσωποι έχουν λάβει τις ε, επιστολές της εκπροσώπησης που είχαμε συμφωνήσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Επειδή είναι πολύ πιεστικό το πρόγραμμά μας, θα έλεγα να περάσουμε αμέσω στο πρώτο σημείο χωρίς καθυστερήσεις. Για το υπόλοιπο της ημερήσιας διάταξης θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συμπρόεδρό μου από το Αυστριακό Κοινοβούλιο, στην Άγγελα Λούικερ. Αξιότιμη κύριε Μωράες, σας ευχαριστώ για τα καλά σας εισαγωγικά λόγια. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο των Κρατών Μελών. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στην ε, συνεδρίαση αυτή της Μεκτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ευρωπόλ και έχω την ευκαιρία να συμπροεδρεύω με τον πρόεδρο της Επιτροπής Λίβε Μωράες. Μέχρι τώρα το όργανο αυτό έχει συνεδριάσει και έχει ασχοληθεί κυρίως με θέματα διαδικαστικά, με τον ειδικό του κανονισμό. Στη Σόφια λύθηκε αυτό στην τελευταία συνεδρίαση και τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε και να συγκεντρωθούμε στο ουσιαστικό μας έργο που είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ. Η οργάνωση αυτή, η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει ε, αποκτήσει μεγάλη σημασία. Ε, το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και ε, μάλιστα υπάρχουν και ε, δίκτυα που χρησιμοποιούν πολλές φορές τις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες για να διευρύνουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Ε, έγκλημα διακίνηση ανθρώπων, τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα. Είναι λίγα από τα εγκλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτικέ αρχές. Η Ευρωπόλ έχει ιδιαίτερη θέση και παίζει ιδιαίτερο όσο και αποφασιστικό ρόλο στα θέματα αυτά. Υποστηρικτικό προς τις διοκτικές αρχές των κρατών μελών. Τι επόμενες ώρες, το επόμενο διήμερο, θα ασχοληθούμε με τις διάφορους τομείς δραστηριοτήτων και πεπραγμένων της ε, Ευρωπόλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριες και κύριοι, επειδή είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη, θα πρότεινα να περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο. Ε, Ποιο θέλει το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Κανείς από ό,τι βλέπω. So, Και θα ξαναδώσω την Προεδρία στον Πρόεδρο. Okay, thank you, Angela. So now... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγγελα. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. For this next point. Γι' αυτό λοιπόν θα προσκαλέσω στο Προεδρείο τους ομιλητές. Παρακαλώ ελάτε να καθίσετε εδώ. ο εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Στρετάνοφ, ο κύριος Βάιτιγκερ, η κυρία Φλωρέα. Παρακαλώ ελάτε στο Προεδρείο αν θέλετε. Και θα σας παρουσιάσω το σημείο. Όπως είχαμε ε, συμφωνήσει στη Σόφια τον περασμένο Μάρτιο, η έννοια της προεδρικής τρόικας, της τρόικας των Προεδριών, έχει ε, συμπεριληφθεί στον ε, εσωτερικό μας κανονισμό μάλλον στο, στους κανόνες διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η, η Τρόικα των Προεδριών αποτελείται από τους επικεφαλής αντιπροσωπιών των πρώην τρεχουσών και μελλοντικών ε, προεδριών του Κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Θέλουμε λοιπόν να ανεπτυχθεί κι άλλο αυτό το σώμα και να προωθήσουμε τις ε, εργασίες μας. Γι' αυτό ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ, η DPS και ο πρόεδρος του Δικητικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν από την επόμενη φορά σε κάθε συνεδρίαση. Ελπίζουμε αυτή η μόνιμη πρόσκληση ε, στις ε, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει αποδεκτή βάσει του πνεύματος του κανονισμού της Ευρωπόλ. Και επίσης ε, τα αιτήματά μας προς τη γραμματεία της ΜΟΚΕ ελπίζουμε να αποστέλλονται εγκαίρω όπω θα πρέπει να γίνει στο Βουκουρέστι τον Φεβρουάριο. Θα, θα καλέσω τώρα του ομιλητέ μα να μα μιλήσουν για τι προτεραιότητε τη ΜΟΚΕ και Άγγελα, παρακαλώ να δώσω το λόγο στου επιμέρου ομιλητέ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Τσβέταν Τσβετάνοφ, πρόεδρο Επιτροπή Εσωτερική Ασφάλεια και Δημόσια Τάξη τη 44η ε, Εθνοσυνέλευση τη Βουλγαρική Δημοκρατία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Уважаеми съпредседатели от Κυρίες και κύριοι, Αγαπητή κυρία Κατρίν Ντεμπόλ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας ε, εδώ. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της Βουλγάρικης Προεδρίας και της δραστηριότητας της ε, Τρόικας των Προεδριών. Ε, Βουλγαρία, Ρωμανία, Αυστρία. Μία από τις προτεραιότητες ήταν η σταθερότητα και η ασφάλεια. Εργαστήκαμε στεναρά πάνω στα θέματα ασφάλειας, ε, ε, πολιτική ασύλου, μεταναστευτικό, μια ισορροπημένη προσέγγιση και ε, οι πηγές της μετανάστευσης, ε, αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, συνεργασία ανάμεσα στα, στους διάφορους φορείς. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, πρόοδο στους διάφορους τομείς. Έχουμε επιτύχει ε, συμφωνία για τα, ε, τις, τους τρεις κανονισμούς του συστήματος ενημέρωσης ε, Σέγγεν. Έχουμε ολοκληρώσει τις συζητήσεις για τη διεύρυνση των εξουσιών της Γιουρολίζα. Έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για το κανονισμό για το νέο σύστημα αιτίας έχουμε επιτύχει μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο για τους δύο κανονισμούς, για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων ενημέρωσης και το νέο πολιτικό κύκλο για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εργασιών. Έχουν ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η προσθέμενη αξία αυτού του συστήματος στα πλαίσια του νέου κύκλου. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ορατότητα των μέσων για την αντιμετώπιση του ε, εγκλήματος. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, έχει υποστεί αξιολόγηση. Κάναμε μια ευρεία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. εξετάσαμε τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ και την προστιθέμενη αξία ε, της Ευρωπόλ το θέμα θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα για τη Βουλγαρία, η εφαρμογή των αποφάσεων της ε, ΜΟΚΕ, η σταθερότητα πολιτική και γεωγραφική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την κατάσταση στα Βαλκάνια. Γι' αυτό και ε, επρόκειτο για προτεραιότητα των ε, συνεδριάσεων μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν τη βάση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τη συνέχεια ε, στις ε, αξίες που έχει προβάλει η Αυστριακή Προεδρία. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι προτεραιότητες θα συνεχίσουν να προβάλλονται και από τη νέα Προεδρία και από τις, ε, την Προεδρία της Αυστρίας και από αυτήν της ε, Ρουμανίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσβετάνοφ. Και τώρα το λόγο έχει ο Αυστριακός συνάδελφος Πέτερ Βάιντιγκερ που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Κάτω Βουλής της Αυστρίας. Danke. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, ω εκπρόσωπο τη Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια σαφή διαπίστωση. Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις ε, στον τομέα της ασφάλειας. Από τη μια, η κρίση ασφαλείας έχει σχέση με μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων από τον Ιανουάριο του 2016 και έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται πολύ πιο στενά από ό,τι μέχρι σήμερα ε, σε ό,τι αφορά τις απειλές ασφαλείας, πόσο μάλλον που το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτο. Από την άλλη, είχαμε και την κρίση του μεταναστευτικού από το 2015 που έδειξε ότι το Σέγγεν και η ελευθερία των ταξιδίων στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνται δεδομένα και αυτονόητα. Χωρί όμω αποτελεσματική προστασία των συνόρων τίθενται θέματα και για την εσωτερική ασφάλεια. Υπάρχουν προκλήσεις λοιπόν με τη μετανάστευση και την ολοκλήρωση στον τομέα της ασφάλειας, πράγμα που παρέβλεπε μέχρι τώρα για πολύ καιρό η Ευρώπη. Η Αυστριακή Προεδρία λοιπόν σήμερα ε, λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ επίκαιρο περιβάλλον. Το στοιχείο της ασφάλειας είναι για μας το κεντρικό ζήτημα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σωστά περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εξού και ε, το πρόγραμμα της Προεδρίας μας είναι υπό το σύνθημα «Μια Ευρώπη που προστατεύει». Δύο ε, κέντρα βάρους της Αυστριακής Προεδρίας έρχονται να συγκεκριμενοποιήσουν το σύνθημα αυτό. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ασφάλεια και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και το φέρνει στο προσκήνιο. Θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών δυνατοτήτων επιστροφής. Αυτό κυριάρχησε ω θέμα και στην άτυπη σύνοδο κορυφή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Σάλτσμπουργκ στις 19 και 20 του μηνός Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο κέντρο βάρου είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα στη γειτονία μα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Η περιοχή αυτή που είναι στην άμεση γειτονία μας έχει τεράστια σημασία όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Μια σαφής προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερη σημασία και πολύ ουσιαστική για τις χώρες αυτές. Το 2018 είναι αποφασιστική χρονιά για ολόκληρη την περιφέρεια εκεί. Μια πολιτική ε, κίνηση και ένα έναυσμα για ε, το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν απαραίτητα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ασφάλεια και η ειρήνη στην Ευρώπη είναι δυνατές μόνο ε, εάν στην άμεση γειτονία μας ε, κυριαρχούν σταθερότητα και ασφάλεια. Και η Ευρωπόλ ως διοκτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κυρίες και κύριοι σαφή στόχο να κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη. Ένα στόχο από τον οποίο όλοι οι πολίτες της Ένωσης εποφελούνται. Είναι μεγάλη απειλή τα μεγάλα εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα, απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για την ασφάλεια και την ίδια την ύπαρξη των πολιτών μας. Η Ευρωπόλ στην καταπολέμηση αυτών των απειλών ε, έχει σαφείς προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Αυστριακή Σκοπιά. Εκτός από όσα σας είπα για την ανάπτυξη των σχέσεων μας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να έχουμε και ένα επιμερισμό των υποχρεώσεων και των καθηκόντων και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνεροφυλακή και Ακτοφυλακή Frontex. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα πρώτο βήμα είναι η πρώτη καινή συνεδρίαση των διοικητικών μας συμβουλίων, των συμβουλίων των δύο μάλλον οργανισμών, στις 4 Οκτωβρίου του 2018. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις συνέργειες και να τις αξιοποιήσουμε. Άλλη προτεραιότητα, συνεργασία στα πλαίσια της παράτυπης ε, μετανάστευσης. Για το λόγο αυτό η Αυστρία έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πλατφόρμα Impact ε, για την καταπολέμηση της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι για την καταπολέμηση της διακίνησης και του λεμπορίου στη Βαλκανική Οδό ε, ε, η Αυστριακή αστυνομία έχει δημιουργήσει ένα διεθνές κοινό επιχειρησιακό γραφείο για να έχουμε πιο γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ και ε, να επιταχύνονται οι διαδικασίες σε περίπτωση διώξεων τέτοιων ομάδων. Άλλα σημαντικά στοιχεία που απασχολούν το impact είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, ε, λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη ε, διάδοση πυροβόλων όπλων χειρός, ε, οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με την περιουσία, περιβαλλοντικό έγκλημα και διάφορα οικονομικά εγκλήματα, Όπω είναι απάτη, πλαστογραφία μέσων πληρωμών, ξέπλυμα χρήματο και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προϊόντων εγκλήματο. Σε αυτά τα βασικά σημεία θα πρέπει να έχουμε απτέ και χειροπιαστέ πρόοδος. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ πάντα σε σχέση με τι προτεραιότητε τη Αυστριακή Προεδρία στο εξή σημαντικό, που είναι ιδιαίτερο μέλημα τη Προεδρία μα. Αυτό είναι ο προπολογισμό της Ευρωπόλ για το 2019. Εδώ οι διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Ευρωπόλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία, ούτε είναι ικανοποιητικέ. Το πλαίσιο που ζητάει η Ευρωπόλ δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη οι προσκεκλημένοι εξωματικοί guest officer της ε, Ευρωπόλ στην Ιταλία και στην Ελλάδα δεν έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί Μάλλον δεν μπόρεσαν να αναβαθμιστούν τα συστήματα πληροφορική και επικοινωνιών τη Ευρωπόλ λόγω έλλειψη χρημάτων. Και δυστυχώ φοβούμαι ότι και το 19 δεν θα συμβεί αυτό. Μιλώντα με εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, συμφωνήσαμε ότι χρειάζονται αυξήσει σε τρία βασικά σημεία. Αυτό όμω δεν πέρασε στην τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια γιατί δεν βρήκε την απαραίτητη πλειοψηφία. Αν θέλουμε όμω να παίρνουμε σοβαρά την καταπολέμηση του εγκλήματο και τη ε, τρομοκρατία, θα πρέπει η Ευρωπόλ να έχει τα χρήματα που χρειάζεται. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μα. Κυρίε και κύριοι, η ε, μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ είναι νεοσύστατο όργανο έχει όμως ε, μια ιδιαίτερη θέση και δεσπόζει. Εδώ δεν θα πρέπει να γίνεται μια γενική ε, ανταλλαγή απόψεων και φιλολογική συζήτηση, αλλά ε, ο κανονισμός της Ευρωπόλ δίνει συγκεκριμένη εντολή σε αυτό εδώ το όργανο που είναι ο πολιτικός κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ από δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των λαών. και εξαρτάται και από τον τρόπο συνεργασίας ε, του Διοικητικού Συμβουλίου με ε, το ελεγκτικό όργανο η σωστή λειτουργία της Ευρωπόλ. Θα πρέπει να οικοδομηθεί αμοιβαία κατανόηση και κοινέ πρακτικές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό. Μια επικοδομητική σχέση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΜΟΚΕ είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε και τα δύο όργανα ε, να μπορούν να αναπτύσσουν πλήρω και να ασκούν τις ε, δραστηριότητες τους. Οι εμπειρίε από τις πρώτες συνεδριάσεις είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι στα πλαίσια μια μιας όσο και επικοδομητική συνεργασίας με την κοινή ανάλυση των σημαντικών ερωτημάτων που αφορούν την Ευρωπόλ θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Και ε, χαίρομαι και προσβλέπω στη συνέχεια των σημερινών συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάιντιγκερ και τώρα η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Οάννα Κονσουέλα Φλωρέα, μέλος της Βουλής και της κοινή Επιτροπής Βουλής και Γερουσίας για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων των Ρουμανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. SRE. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Φλουρέ. Thank you. Ευχαριστώ. Πριν σας πω κάποια σχόλια για τις προτεραιότητές μας για το 2019, να ευχαριστήσω τους συμπροέδρους μας. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την συνάντηση θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσβετάνοφ από τη Βουλγαρία και από το Ευρωκοινοβούλιο τον κύριο Μωράης για τις προσπάθειές τους ε, και από τη Σόφια. Τώρα έχουμε έναν ιστορικό κανονισμό και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας με κάποια ε, συνοχή. Θα συνεχίσω στη γλώσσα μου. νόστρου πριντσιπάλ, ον βασικός μας στόχος ε, στο πλαίσιο της Τρόικας των Πέτριών είναι να θέσουμε στο κέντρο των συζητήσεων στα ζωτικότερα θέματα για την ομάδα αυτή. Υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το υπάρχον πλαίσιο και θα κάνουμε επικοδομητικές συνεισφορές όπου αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι ο χρόνος και η εμπειρία θα μας δείξουν αν έχουμε καταφέρει σωστά αποτελέσματα. Για να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες για το πρώτο εξάμεινο του 2018, θα φανούμε διαλλακτικοί και ευέλικτοι, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις. Όμως ήδη πρέπει να σκεφτούμε ότι στο κέντρο των προτεραιοτήτων μας πρέπει να βρίσκονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να καταλαβαίνουν και να κατανοούν γιατί οι δράσεις της Ευρωπόλ είναι τόσο σημαντικές και κατά ποιον τρόπο τα δικαιώματά τους, οι ελευθερίες τους, οι δικές μας αξίες και αρχές προωθούνται. Ε, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο συνεργασία των κατών μελών κατά της τρομοκρατίας, κατά των κυβέρνων επιθέσεων που είναι διασυνοριακού χαρακτήρα αυτού του είδους το συντονισμό θέλουμε για να εδραιώσουμε το ρόλο και την σημασία της Ευρωπόλ ως ένα κομβικό σημείο συγκέντρωσης πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε και την απαραίτητη υποστήριξη, ποιοτική υποστήριξη στις έρευνες που διοργανώνονται στα εθνικά κράτη-μέλη. Η ποιότητα των πληροφοριών που αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο ε, και η ταχεία απόκριση, ε, η προσφορά απαντήσεων όταν τίθενται ερωτήματα, είναι απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας που έχουμε διοργανώσει με τα κάτι μελη ε, μιλάμε για συνεργασία έντονη και εντατική, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα σύνορα και να μπορούμε να διαχειριστούμε τις απειλές και τους κινδύνους κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της λαθρομετανάστευσης. Επίσης κατά της ριζοσπαστικοποίησης. και αν μη τι άλλο για έναν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για το 2019-2021. Κυρίε και κύριοι, το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση των παραβιάσεων και παρανομιών στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι έχουμε περίπου 70 ε, ειδικού, ε, ειδικού της πληροφορική κυρίω, που ήδη ε, έχουν προσληφθεί και εργάζονται σε αυτό το σώμα. Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, αυτούς τους τελευταίους μήνες, στη μετανάστευση, στην πολιτική ασύλου, στις εσωτερικές υποθέσεις της Ένωσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα θέματα. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή από πλευρά μα και να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατία θα είναι επίσης μια από τις βασικές προτεραιότητε για το πρώτο εξάμεινο του 2019 δεδομένη τη στρατηγικής για τις εξωτερικές υποθέσει της Ευρωπόλ για το 2019-2021 πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον να έχει προεξάρχοντα ρόλο ό,τι αφορά την ασφάλεια σε, παγκόσμιο, σε παγκόσμια κλίματα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και αυτό συνάδηκε με την αντίληψη που είχαν διαμορφώσει οι προηγούμενες τρόικες προεδριών. Η ανατολική γειτονία, η πολιτική μας για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι κεντρική σημασία για την πολιτική μας ατζέντα. Φίλες και φίλοι, οι ερχόμενες ευρωεκλογέ φέρνουν τους Ευρωπαίους πολίτες στο κέντρο όλων μα των μεριμνών και των προσπαθειών ε, είναι σαφές ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις δικές τους προσδοκίες, στις δικές τους ανάγκες. Διότι η τρομοκρατική απειλή συνεχίζει να τους βαραίνει. Είναι ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα ασφάλειας που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να είναι μια υποχρέωση για το κάθε κράτος με μέλος μεμονωμένα, αλλά πρέπει να γίνει μια ευθύνη συλλογική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφάλεια είναι ο κεντρικός πυλώνας της Ρουμανικής Προεδρίας. Θα φροντίσουμε να το συζητήσουμε ε, σε πολλές ε, περιστάσεις. Θα οργανώσουμε τέτοιες συζητήσεις συστηματικά. Και ελπίζουμε στη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας περιμένω από το Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φλωρέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και τους τρεις ομιλητές της Τρόικα, των τριών διαδοχικών προεδριών. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μερισσές διάταξης, που είναι ε, ο πολιετής προγραμματισμός ε, της Ευρωπόλ. Το αντίστοιχο σχέδιο έχει αποσταλεί ε, στις 7 Ιανουαρίου σε όλες τις αντιπροσωπείες προς εξέταση. Στη Σόφια στη συνέχεια κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και οι διάφορες αντιπροσωπείες είχαν ευκαιρία μέχρι τις 29 Αυγούστου να υποβάλουν γραπτός τις προτάσεις τους στη γραμματεία της ΜΟΚΕ. Έχουμε λάβει γραπτές τοποθετήσεις από την Κυπριακή και τη Ρουμανική Αντιπροσωπεία. Πριν δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ντεμπόλ για να μας κάνει μια εισαγωγή, θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση και πώς θα διαρθρωθεί αυτή για το επόμενο θέμα. Έχουμε την εξής φόρμουλα. Εναλλάξ θα παίρνουν το λόγο δύο εκπρόσωποι από Εθνικά Κοινοβούλια και ένα μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Γιατί οι πρόσωποι ε, που θέλουν το λόγο παρακαλούνται να συμπληρώνουν ε, την αντίστοιχη καρτέλα ε, με το θέμα της ημερήσιας διάταξης και να τα δίνουν στη γραμματεία για να τα φέρνει στο Προεδρείο. Ο κατάλογος των ομιλητών θα καταρτιστεί με βάση τις κάρτες που θα πάρουμε και με τη σειρά που θα φτάνουν στο Προεδρείο. Και θέλω να πω ότι και οι εκπρόσωποι από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου έχουν τέτοιες κάρτες ε, και πρέπει να τις συμπληρώσουν ανάλογα με το χρώμα αν θέλουν το λόγο για ένα θέμα της μέρης της διάταξης. Λοιπόν, προτείνω και χρόνο αγόρευσης να περιοριστεί στο δίλεπτο αναομιλητή. Επιφυλάσσομαι όμως, ανάλογα με τον αριθμό των παρεμβάσεων, να προσαρμόσω και το χρόνο αγόρευσης, έτσι ώστε όλοι να πάρουν το λόγο, όλοι όσοι το επιθυμούν και το έχουν δηλώσει. Παρακαλώ την εκτελεστική διευθύντρια κυρία Ντεμπόλ να σκάνει την εισαγωγική της δεκάλεπτη παρουσίαση. Παρακαλώ και ε, μετά ακολουθεί η συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Distinguished members. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές των εθνικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μωρά, κυρία Λιγκέρ, Ευχαριστώ που με προσκαλείτε εδώ ε, στην τρίτη συνεδρίαση της Μεκτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και είναι η πρώτη φορά υπό την ιδιότητά μου ως εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπόλη. Στην προηγούμενη συνεδρίασή σας τον Απρίλιο ήμουν εδώ ως παρατηρήτρια και πρέπει να πω ότι έφυγα από τη συνεδρίαση με πολύ θετικά συναισθήματα. Ήμουν βεβαία ότι η ΜΟΚΕ θα ενισχύσει την Ευρωπόλ και την αξιοπιστία μας αλλά και την νομιμοποίησή μα ενώπιον των πολιτών. Εσεί, η μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, προσδίδετε στην Ευρωπόλ ε, μια άλλη ε, δυνατότητα ε, να έρθει πιο κοντά στου Ευρωπαίου πολίτε, ξεφεύγοντα από το στενό πλαίσιο αρμοδιοτήτων τη. Έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου εδώ και πέντε μήνε και στο τρίτο μήνα ε, δουλειά μου στην ε, Επιτροπή Λίμπε τη 9 Ιουλίου τόνισα ότι η Ευρωπόλ είναι ένα εύρωστο οργανισμό, λειτουργεί εύρυθμα και ότι στόχο μου είναι να γίνει ακόμα ισχυρότερο. Όμω συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη. Μπορώ να το κάνω μόνο με τη στήριξη όλων των ε, συμμετεχόντων και ενδιαφερομένων. Ω εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μελετήσω τις ανάγκες και τις μέρημνε όλων των συμμετεχόντων και των ε, ενδιαφερομένων. Οι τελικοί καταναλωτέ είναι οι ιδιοκτικέ αρχέ των κρατών μελών. Ε, γι' αυτό αποφάσισα να συναντήσω όλους τους επικεφαλείς αστυνομίας και διοκτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αφιέρωσα κάποιες μέρες σε επισκέψεις προς αυτούς για να μιλήσουμε για τις προσδοκίες τους σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, επιτόπου. Οι επισκέψεις αυτές μου δώσαν τη δυνατότητα να διαμορφώσω εικόνα για να ενισχύσω και να βελτιώσω τη στήριξη που προσφέρει η Ευρωπόλη στις εθνικές αρχές. Η ανταπόκριση που είχα από του επικεφαλεί αστυνομία ήταν καλή. Έλαβα την επιβεβαίωση ότι η Ευρωπόλ είναι ένα εύρυθμα λειτουργών οργανισμό. Οι εθνικέ διοκτικέ αρχέ ε, εκτιμούν και ευχαριστούν την Ευρωπόλ για την προσφορά τη, ιδίω στον, στον εγκληματικότητα του κυβερνοχώρου, την ε, τρομοκρατία και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Οι εθνικέ αρχέ όμω θέλουν περισσότερα Θέλουν περισσότερα από την Ευρωπόλ για να είναι επιτυχή η καταπολέμηση του διεθνού οργανωμένου εγκλήματο και τη τρομοκρατία. Θέλουν περισσότερη στήριξη. Θέλουν περισσότερη στήριξη στην καταπολέμηση τη διακίνηση ναρκωτικών, τη δίωξη οικονομικού εγκλήματο και του κύβερνου εγκλήματο συγκεκριμένο αίτημα έχει απευθυνθεί προ την Ευρωπόλ για να ενισχυθούν οι δυνατότητε ανάλυση δεδομένων για να υποστηρίξουμε καλύτερα και να αποθάλψουμε καλύτερα τι έρευνε των κρατών μελών. Η Ευρωπόλ ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία αυτή και α, ήδη μελετάμε τα κράτη-μέλη πώ μπορούν οι ε, υπηρεσίε ανάλυση δεδομένων τη Ευρωπόλ και των εθνικών κρατών να ενισχυθούν. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι να τυποποιήσει την ε, ανάλυση δεδομένων που έχουν σχέση με παράνομες ενέργειες και έγκλημα ε, για να εντοπίζουμε πιο εύκολα υπόπτους αλλά και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή ε, ειδικών τεχνικών πληροφοριών που προκύπτουν από ανάλυση. Επίσης θα προβλέψουμε κοινή εκπαίδευση των ε, επεξεργαστών πληροφοριών σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι διοκτικέ αρχέ και οι επικεφαλεί αστυνομία θέλουν να είναι έτοιμοι για τα δεδομένα του αύριο. Ελπίζουν ότι η Ευρωπόλ θα του υποστηρίξει στη διαχείριση και την ε, ανάλυση των μεγάλων δεδομένων. Οι επικεφαλεί από τα κράτη-μέλη περιμένουν η Ευρωπόλ να γίνει ένα κομβικό σημείο της καινοτομία και της ψηφιοποίηση τη αστυνομική δράση καθώς και ανταλλαγής τεχνικών ε, γνώσεων. Οι επικεφαλεί επίσης ζήτησαν να υπάρχει ακόμη περισσότερη επιχειρησιακή ε, προσπάθεια με στόχο τα αποτελέσματα. Αυτό θα κάνουμε το 2019 σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις διοκτικές τους αρχές θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να ενισχυθούμε και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλω να ευχαριστήσω ήδη τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και Κιν και τη Γενική Διεύθυνση Home, η οποία έχει ειδική σημασία για μας ε, και την, ε, τον οργανισμό μας και θα φροντίσουμε την καλή σχέση εμπιστοσύνη που έχουμε να την ε, ε, προωθήσουμε και στο μέλλον. Οι αποδείξει που έχουμε και τα δεδομένα για το, για το έγκλημα στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χρήσιμα για την Ευρωπόλη και τα καλωσορίζουμε. Μια ακόμα προτεραιότητα για μένα είναι να ενισχυθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του διεθνεί οργανισμού στους πέντε μήνες ε, άσκησης των καθηκόντων μου έχω συναντήσει τους εκτελεστικούς διευθυντές της Ευρωπαϊκής Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής, της ε, Eurojust, της EULISA, ε, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του, του Οργανισμού Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών, της του Οργανισμού για τον Καταπολέμηση των Χημικών Όπλων και ούτω καθεξής. Ε, στο επίπεδο του οργανισμού μας την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και κοινό, ε, κοινή συνεδρία του Διοικητικό Συμβουλίου για να συζητήσουμε ε, κάποια εκκρεμή ζητήματα. Θέλω η, Ευρωπα... η Ευρωπόλ να γίνει κινητήριος δύναμη αυτών των κοινών προσπαθειών και μόνο με ε, ισχυρά δίκτυα θα έχουμε στενή συνεργασία. μόνο αν έχουμε ανταλλαγή ειδικών γνώσεων και πληροφοριών με τους υπόλοιπους οργανισμούς θα καλύψουμε το χάσμα των μυστικών και ειδικών πληροφοριών και θα γίνουμε ισχυρότεροι. Από τις απαντήσεις που έλαβα από τις εθνικές αρχές πολύ χρήσιμα πορίσματα, τα οποία θα συζητηθούν την Τετάρτη και Πέμπτη στην ε, Σύνοδο των ε, ε, Αστυνομικών Διευθυντών στην Χάγη, το μεγαλύτερη εκδήλωση που οργανώνει η Ευρωπόλ. Στην συνάντηση αυτή θα καταρτήσουμε και τη στρατηγική για τον οργανισμό μα. Για να ολοκληρώσω, το πρώτο πεντάμινο δουλειά μου ήταν πολύ επιτυχέ. Η Ευρωπόλ υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη στι δράσει τη. Έμαθα πολλά για του οργανισμού και τι ανάγκε των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μα. Είμαι ότι τα θεμέλια για το μέλλον ε, που έχει ήδη θέσει η Ευρωπόλ ε, θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Ε, θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε το έγγραφο για τον πολιετή προγραμματισμό 2019-2021 όπου ένα πρώτο σχέδιο του εγγράφου έχει ήδη υποβληθεί από τον Μάρτιο στην ε, συνεδρίαση που προείδρευε ακόμα ο Ρόμπ Βέινραϊτ. Δεν έχουν γίνει αλλαγέ έκτοτε από τον Μάρτιο και η τελική έγκριση προβλέπεται θα τέλη Νοεμβρίου. Στο έγγραφο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι τη Ευρωπόλ αναφέρονται ξεκάθαρα. Πρώτος στρατηγικός στόχος είναι η Ευρωπόλ να γίνει κομβικό κέντρο συγκέντρωσης ε, πληροφοριών για το έγκλημα και ε, να αποστέλλονται αυτές οι ειδικές γνώσεις σε όσους τα χρειάζονται στα κράτη-μέλη. Επίσης, ως προς την πληροφόρηση και τη διαχείριση των πληροφοριών, θα αξιοποιήσουμε νέες δυνατότητες για να βελτιώσουμε το τοπίο των μυστικών πληροφοριών και της ανάλυσης τους ε, στα κράτη-μέλη. Η κοινή διαχείριση δεδομένων θα συνεχιστεί ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πολλοί επικεφαλεί αστυνομιών και αστυνομικοί διευθυντέ μου είπαν στι επισκέψει μου ότι επενδύουν στη διαχείριση των δεδομένων. Στην Ευρωπόλη ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά μα επικεντρώνεται στον τομέα τη πληροφορική. Κοιτάζουμε να ετοιμάσουμε τα συστήματά μα ώστε να είναι διαλειτουργικά και να μπορούν να συνδυαστούν με άλλα συστήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φροντίσουμε να δούμε πώς μπορούμε ας πούμε, να ενσωματώσουμε το ΣΥΣ2. Αυτό βέβαια απορροφά ένα μέρος του προπολογισμού μας αρκετά μεγάλο. Όμως είναι σημαντικό τα συστήματά μας να είναι πλήρως επικυρωποιημένα και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέα εργαλεία. Ε, ο επόμενος στρατηγικός στόχος έχει να κάνει με το να μπορεί η Ευρωπόλη να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη και πυρογνωμοσύνη για τις έρευνες των κατώμελών. Προηγουμένως έκανα λόγο για τις προσδοκίες των κατώμελών στα επιχειρησιακά και πώς μπορώ εγώ να απαντήσω στις ε, ανάγκες που εξέφρασαν οι εθνικές αρχές. Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στην Σύνοδο των Αστυνομικών Διευθυντών στη Χάγη αυτή την εβδομάδα. Εδώ λοιπόν ε, η Ευρωπόλ θέλει να είναι ένας αποτελεσματικός οργανισμός με αποτελεσματική διοργάνωση. Το 2017 η Ευρωπόλ ε, διαχειρίστηκε έναν προπολογισμό 114,6 εκατομμυρίων και πέτυχε 80% ε, καλής απορρόφησης των κονδυλίων. Αυτό έχει, δείχνει τη σημασία της, ε, του προπολογισμού της Ευρωπόλ για το 2019 και τα επόμενα χρόνια και στα, στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δυστυχώς η τωρινή πρόταση για την Ευρωπόλ και για το 2019 είναι χαμηλότερη από τις προσδοκίες μας και από τις πραγματικές ανάγκες της Ευρωπόλ. Μάλιστα επιβάλλει μεγάλη μείωση σε σχέση με το, τον προπολογισμό του 2018. Ε, υπολογίζουμε στην ε, υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καλυφθεί αυτό το κενό Στι προφορίες που θα έχετε στην Επιτροπή Προπολογισμού αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε σε συνεννόηση με τι εθνικέ σα κυβερνήσει και με ευαισθητοποίηση στα δικά μα θέματα σε εθνικό επίπεδο να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσει. Η συνεργασία με, άλλες, ε, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης είναι επίση σημαντικό. Θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα αλλά και διαλεκτικότητα στο να μπορέσει η διαθεσμική συνεργασία να γίνει πιο πλαισιωμένη, στοχευμένη και αποτελεσματική Συζητήσαμε με όλου του οργανισμού που μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μα σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. Ε, πέραν του δικτύου ε, για την, των οργανισμών καταπολέμησης του εγκλήματος από το 2018 θα συνεχίσουμε την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας για να δούμε τι σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε. Πρωτού ολοκληρώσω να σημειώσω την στήριξη που προσφέραμε στις έρευνες στην ε, Μάλτα και τη Δημοκρατία της Σλοβακίας. Τον περασμένο χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο επικεντρώθηκε στην τήρηση του κράτους δικαίου και την προστασία του για το πόσο σημασία έχουν τέτοιου είδους έρευνες. Η Ευρωπόλ θα συνεχίσει να στηρίζει τις αρχές της Μάλτας και της Σλοβακίας στις ερευνητικές τους προσπάθειες. Όπως και στο παρελθόν δεν θα αναπαυθούμε στις δάφνες μας και θα φροντίσουμε να επιδιώκουμε διαρκώς την ε, ικανοποίηση των προσδοκιών των κατών και την ε, ε, νέα έκφραση των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα, μάλλον σύντομα, θα συναντηθούμε με μέλη της GPSD και ενθαρρύνω όλους σας να επισκεφθείτε το επιτελείο, το στατηγείο της Ευρωπόλ για να δείτε από κοντά τι συζητήσεις κάνουμε και τι δουλειά ε, και πώς είμαστε οργανωμένοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας απευθυνθώ σήμερα και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Um, και τώρα Συνάδελφοι, αρχίζει η συζήτηση. Νομίζω ότι πρώτοι θα πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι από τη Ρουμανία και την Κύπρο. Sorry, I was getting some... Α, συγγνώμη. Άκουγα Ολλανδικά στα ακουστικά μου, λέει ο Πρόεδρος. Δεν πειράζει. Μπλέξαν οι γραμμές. Λοιπόν, ε, Ρουμανία αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σχολιάσω κάτι από αυτά που είπε η κυρία Ντεμπόλ. Ε, ήταν πολύ εύστοχη ομιλία σας, αλλά δεν θέλω να αφήσω να περάσει αυτό ε, που είπε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, τη συμμετοχή της ΜΟΚΕ. Το είπα και στην Αυστρία πριν από 15 μέρες στην αντίστοιχη συνεδρίαση ασφαλείας. Αν τα δούμε πολύ αντικειμενικά, πρέπει να ξέρουμε και τι αιτήματα δέχεται η Ευρωπόλ που είναι πολύ μικρή ως οργανισμός σε ό,τι αφορά τους συνδέσμους ε, ε, αξιωματικούς, τα hot spot και τα λοιπά. Ο προπολογισμό δεν προσφέρεται καθόλου για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες και τα αιτήματα. Και πραγματικά θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε η τελεστική διευθύντρια στην ομιλία της. Και παρακαλώ κοιτάξτε αυτό το θέμα πάρα πολύ προσεκτικά στις δικές σας συζητήσεις και συνεδριάσεις στα κράτη-μέλη και στα κοινοβούλια για τα δημοσιονομικά, όπως και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε αμέσως στους ομιλητές μας. Η κυρία Φλωρέα από τη Ρουμανία. And I think we also have For speak. Και, ε, λοιπόν, πρέπει σε αυτές τις κάρτες που σας δείχνω, αν θέλετε το λόγο, να τις συμπληρώσετε και να το... Ζητώ συγγνώμη για τη γραφειοκρατία, αλλά αυτή είναι η διαδικασία συνηθισμένη εδώ. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι και να έχουμε κάθε φορά να μιλάει ένας από το Εθνικό Κοινοβούλιο και μετά ένας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. On the blue form, is that correct? Λοιπόν, η γαλάζια κάρτα, που δεν είναι ακριβώς γαλάζια, ε, είναι μπες λίγο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εμεί τη βαφτίζουμε μπλε. Μην μπερδευτείτε. Γράψτε το όνομά σα αν θέλετε το λόγο για το συγκεκριμένο σημείο στη μέρη διάταξη. Και πού είναι η κυρία Φλωρέα, τη χάσαμε. Μα ε, είναι τόσο χανές το εμικύκλιο, δεν σας βλέπω. Κυρία Φλωρέα, έχετε ερώτηση ή σχόλιο για την κυρία Ντεμπόλ. Σύντομα. Μέχρι δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα την πρόθεση να ζητήσω το λόγο, όμως Ήθελα να σας παρουσιάσω τη ε, συμβολή της, τη της Ρουμανίας ε, συγκριτικά με το έγγραφο προγραμματισμού της Ευρωπόλ. Δεν ξέρω αν μπορώ να λάβω το λόγο σχετικά με αυτό το θέμα. Ναι, ναι, βέβαια. Ε, μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματα που θέλετε στην κυρία Ντεμπόλ. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Διαβάσαμε το σχέδιο ε, του εγγράφου προγραμματισμού που παρουσίασε η κυρία ε, Ντεμπόλ. Είναι πολύ καλά δομημένο, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Θα θέλαμε να προβάλλουμε όμως κάποια θέματα. Η αντιπροσωπεία μας θα ήθελε να τονίσει έναν από τους βασικούς στόχους του σχεδίου του εγγράφου προγραμματισμού ε, πρόκειται για την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπόλ στα κράτη-μέλη στις τρεις ε, προτεραιότητες, δηλαδή τρομοκρατία, έγκλημα, οργανωμένο έγκλημα και ηλεκτρονικό έγκλημα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπόλ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται άμεσα σε επιχειριαστικό επίπεδο για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των κρατών μελών, διαθέτοντας τεχνογνωσία και σε πραγματικό χρόνο στους τομείς στόχους. Υπάρχει επίσης το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Η Αυστριακή Προεδρία ε, έχει ως προτεραιότητα ε, την προστασία, την Ευρώπη που προστατεύει, προβάλλοντας τη διάσταση της ε, ασφάλειας και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για ένα θέμα που θα συνεχίσει να είναι ε, σημαντικό τα ερχόμενα χρόνια. Η Ευρωπόλ πρέπει να μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο καταστρέφοντας ε, τις μεθόδους δράσης των διακινητών ουσιαστικά μέσα από την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου που ε, διαχειρίζεται, που θα διαχειριζόταν την ε, ένομη μετανάστευση. Πιστεύουμε ότι η διάθεση της απαραίτητης τεχνολογίας για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας ε, στην Ευρώπη ε, χρειάζεται την υποστήριξη επιπλέον πόρων. Κύριο καθήκον της Ευρωπόλ είναι η συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών. Άρα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των επιπτώσεων του Brexit στο πολιτές πρόγραμμα της Ευρωπόλου. Κλείνοντας, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι βασιζόμαστε στην Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά την προβολή των πρωτοβουλίων της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα έχουμε και την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ τους ερχόμενους μήνες και αυτό σημαίνει ότι θα ενταθεί η συνεργασία της ε, Ρουμανίας με την Ευρωπόλ και φυσικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όσους εργάζονται για την προβολή των στόχων ε, στα πλαίσια του προγραμματισμού 2019-2021. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλωρέα. Σας παρακαλώ συνάδελφοι ε, που θα πάρετε το λόγο να προσπαθήσετε να τηρείτε το δίλεπτό σας για να προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Ερωτήσεις κάντε παρακαλώ ή σχόλια αλλά σύντομα όσο μπορείτε. Ευχαριστώ κύριε Φλωρέα. Πριν προχωρήσουμε στον πρώτο Ευρωβουλευτή έχουμε την Κυπριακή Αντιπροσωπή. Κύριε Δημητρίου παρακαλώ δύο λεπτά. και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μα άποψη είναι ότι το προσχέδιο πολιετού προγραμματισμού είναι ένα συνεκτικό και καλά δομημένο έγγραφο που περιγράφει με σαφήνεια του στρατηγικού στόχου, όπω η κυρία Ντεπόλ του ανέλησε και προηγουμένω. Ωστόσο, θέλουμε να αναφερθούμε σε μερικά σημεία. Καταρχήν, θεωρούμε ότι η διαφθορά αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει μια σειρά άλλων εγκλημάτων όπως αναφέρεται και στο τελευταίο έγγραφο της αξιολόγησης των απειλών. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η αντιμετώπιση της δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο πολιετούς προγραμματισμού. Η ερώτηση είναι πώς σκοπεύει η Ευρωπόλ να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Κρίνεται χρήσιμη η συμπερίληψη μιας τέτοιας αναφοράς. Τώρα, όσον αφορά το στόχο 1.3 για την στρατηγική ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με εταίρους συνεργασίας. Διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις μεσογειακές χώρες με τις οποίες μια συμφωνία ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων θεωρείται επίγουσα. Η χώρα έχει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, γεγονός που επιδεινώνεται περαιτέρω υπό την τρέχουσα θέση σε ισχύ ενός πολύ αυστηρού συνόλου αντιτρομοκρατικού μέτρου. Επιπλέον, η έκθεση προόδου σχετικά με τον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων για του Τούρκου υπηκόου προβλέπει ρητά ότι η Τουρκία πρέπει να αναθεωρήσει την νομοθεσία και τι πρακτικέ τη για την τρομοκρατία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίω μέσω τη καλύτερη ευθυγράμμιση του ορισμού τη τρομοκρατία. Υπό το πρίσμα αυτό, ο σκοπό τη ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία πριν από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας θέτει υπό αμφιβολία πιστεύουμε το πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της ευρωπόλ και της τουρκίας. κάτι πολύ σημαντικό η τουρκία δεν συνεργάζεται με την κύπρο σε θέματα σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας θέτοντας σε κίνδυνο τη συνολική αποτελεσματικότητα των στόχων της ευρωπόλ. Υπό αυτές τις συνθήκες πιστεύουμε πως η αναβάθμιση και η διεύρυνση του συμβατικού πλαισίου της Ευρωπόλ έναντι αυτής της χώρας στέλνει κατά τη γνώμη μας ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα όσον αφορά την πραγματική σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και ειδικότερα η Ευρωπόλ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Μια τελευταία επισήμανση είναι ότι ενώ η σημασία που αποδίδεται στην καταπολέμηση της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης είναι ευπρόσδεκτη η, η ριζοσπαστικοποίηση που διενεργείται σε χώρους θρησκείας, σε τζαμιά ή σε άλλα ιδρύματα θα πρέπει ίσως να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα σε συνεργασία με το δίκτυο ευαισθητοποίησης για την ριζοσπαστικοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, το δίλεπτο, αν γίνεται να τηρείτε, γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος, για να προλάβουμε και να κάνουμε και ερωτήσεις. Στην κυρία Ντεμπόλ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απευθυνθώ στην ε, Διευθύντρια της Ευρωπόλ να τη συγχαρώ. Σε πέντε μήνες έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά, εντατικότατη και αποτελεσματικότατη. Ε, έχουμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες μας ε, σε εσά για την ασφάλεια. Έχω μερικές ερωτήσεις. Ο πρόεδρος Γιούνκερ την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε σε δύο θέματα που θέλω να σας τα υποβάλω προσκέψη. Πρώτον, να αφαιρείτε γρήγορα ε, ε, από ε, το διαδίκτυο περιεχόμενο που αναφέρεται στην τρομοκρατία. Μπορεί σήμερα να το κάνει αυτό η Ευρωπόλ ε, με αυτή τη νέα πρόκληση με το δυναμικό που έχει το ανθρώπινο και τους οικονομικούς πόρους. Δεύτερον, πάλι ο πρόεδρος Γιούνκερ λέει ότι θα προτείνει να ενισχυθούν οι οργανισμοί Frontex που είναι η φυλακή όπως γνωρίζουμε και το ΕΑΣΟ, το γραφείο. Εμένα με ανησυχεί αυτό, γιατί θα πει να ενισχυθούν. Αυτό θα είναι εις βάρος των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων και ικανοτήτων που έχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Διακίνησης Μεταναστών της Ευρωπόλ. Παρακαλώ να σχολιάσετε αυτά τα δύο ερωτήματα. Ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο. Γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι μόνιμο το πρόβλημα, γνωρίζοντας ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη το ηλεκτρονικό έγκλημα ε, ε, αντιπροσωπεύει το μισό έγκλημα της ε, παράνομης δραστηριότητα. Και μιλάτε για επενδύσεις σε νέα εργαλεία και συμφωνώ. Και συμφωνώ και με τον Πρόεδρο ότι θα πρέπει να σας υποστηρίξουμε και να σας πρικοδοτήσουμε πολύ περισσότερο στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στον προϋπολογισμό σας. Έχετε όμως τους απαραίτητους πόρους, ε, προσωπικό, επιμελητία, ε, τεχνολογία για να αντιμετωπίσετε το ηλεκτρονικό έγκλημα στη διάσταση που έχει πάρει. Και τελευταίο, έχω πολλά, αλλά τι να κάνω, τώρα σταματώ εδώ. Τα δίκτυα ε, και την εθνική νομοθεσία. Θα ε, ε, βελτιώσετε το δίκτυο ή θα αλλάξετε το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ε, για τα οικονομικά, το FUNET, για τα οικονομικά εγκλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Δίας Δεμέρα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και πάλι από τη Γαλλία παρακαλώ. Mes chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημερινό πλαίσιο που σηματοδοτείται από την τρομοκρατία, την ε, αύξηση της μετανάσκευσης ε, η Ευρωπόλ πρέπει να γίνει ο οργανισμός που θα βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τρεις από αυτές. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπόλ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα κράτη-μέλη, να προσφέρει επιχειριασιακή συνδρομή. Αυτή η συνεργασία, η ενίσχυση της συνεργασίας χρειάζεται κυρίως στο επίπεδο της ανταλλαγής των ε, πληροφοριών, η οποία πολλαπλασιάστηκε επί 9 τα τελευταία χρόνια. Όμως το 85% της ανταλλαγής ε, το αναλαμβάνουν ε, λίγες χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, η Ευρωπόλ, έχει μεγαλύτερα περιθώρια για να προσφέρει ε, προσθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να στηρίξει τα εθνικά κοινοβούλια, να αξιολογήσουν τη συμβολή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά το Brexit πρέπει να αποφύγουμε να οδηγήσει σε μία αποδυνάμωση της ασφάλειας. Η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απαραίτητη. Υπάρχουν όμως ερωτήματα σε ό,τι αφορά σχέδια συμφωνιών, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην Ευρωπόλη και τις ε, εποπτικές αρχές τους. Αυτό το θέμα δεν ήταν ξεκάθαρο όταν το αναφέρετε το Μάρτιο. Ε, χρειάζεται μια καταπερίπτωση προσέγγιση. Επίσης, η διαλειτουργικότητα των, συστημάτων, των ευρωπαϊκών συστημάτων ενημέρωσης ε, είναι σημαντικός τομέας και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ε, βασικές προκλήσεις η σύνδεση των βάσεων δεδομένων είναι απαραίτητη. Πρέπει να ενισχυθεί. Η Ευρωπόλ πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να έχει πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών προστατεύοντας την, τα προσωπικά δεδομένα. Η διαλειτουργικότητα που προβλέπεται, που προσδοκάται στο 2019-2021 χρειάζεται με ένα νέο προσωταλισμό των πόρων της Ευρωπόλ. Τέλος, η ασφάλεια στο κυβερνοχώρο αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Η Ευρωπόλ το θεωρεί ε, προτεραιότητα αυτό το θέμα και το χαίρομαι γι' αυτό. το ηλεκτρονικό έγκλημα αποτελεί αυξανόμενη απειλή με σοβαρές επιπτώσεις. Χρειαζόμαστε μια ολική προσέγγιση και στενή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες επιβαλής του νόμου ε, της Ευρώπης καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα και με τον τραπεζικό τομέα ιδιαίτερα. Αυτές είναι για μένα να κάποιες από τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να ε, ενταχθούν στην στον πολιετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ και χαίρομαι που οι συνάδελφοι από τη Ρουμανία και την Κύπρο μοιράζονται αυτές τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε να πω ότι δύο πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρευρίσκονται ο Λόρδος Κέρκοπ, Τίμωθη Κέρκοπ, καλώς όρισες Τίμωθη, και η κυρία Ρία Όμεν Ράιτεν. Καλώς ορίσατε θερμότατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δυο σας. Από τη Βουλγαρία τώρα ο κύριος Τσβετάνοφ, παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να σχολιάσω το έγγραφο προγραμματισμού. Πράγματι, είναι σωστό να ορίζουμε σε διετία, σε αυτή τη διετία την πρόπτικη εξέλιξη του οργανισμού ω προ τι δυνατότητέ τη, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ώστε πραγματικά να μπορεί να υποστηρίξει τι επιχειρησιακέ δράσει και τι έρευνε των 100 Δύο στοιχεία θέλω να σχολιάσω, τη στρατηγική και του απαραίτητου πόρους, τα κονδύλια δηλαδή, για την ε, υλοποίηση της στρατηγική αυτής. Πρέπει να πρικοδοτήσουμε επαρκώ την Ευρωπόλ για να μπορεί να λειτουργεί ε, αποτελεσματικά. Καλώς ε, προσπαθήσαμε να επικεντρώσουμε αρκετά κονδύλια στην καινοτομία και τους πόρους της πληροφορικής. Όμως πρέπει να δούμε τι πόρους απαιτεί και η μεταναστευτική κρίση με τις πιέσεις που ασκεί και οι ενδεχόμενες τρομοκρατικές απειλές. Ως προς την ε, διάσταση αυτή λοιπόν καλωσορίζω την πρωτοβουλία του οργανισμού να συνεχίσει να ε, προωθεί τη δράση της στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις συμφωνίες με τους υπάρχοντες μηχανισμούς συνεργασίας διότι υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να παραμείνουν κοντά στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στη δράση της Ευρωπόλ και να παραμείνουν πιστές στην κοινή ερμηνεία των αξιών αυτών. Αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε ένα κενό πολιτικών αξιών και ελευθεριών στην ευρύτερη περιοχή και θα μπορέσουν και οι πολίτες της χώρας να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές προκλήσεις που, τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Ε, τώρα για την μετανάστευση και τις πιέσεις που ασκούνται στις κοινωνίες μας είναι σημαντικό η Ευρωπόλη να λάβει υπόψη και το ρόλο της Τουρκίας σε αυτό το θέμα ε, και να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή. Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό θέμα, το Brexit. Υπάρχουν μεταναστευτικές ροές που επιστρέφονται στην Τουρκία αντί να προωθούνται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Και ε, να ξανάρθω στο Brexit. Ε, το Brexit είναι ένα ε, στυλοβάτη, ένα πυλώνα τη ασφάλεια μα. Τι θα κάνουμε για να διατηρήσουμε του μηχανισμού που μα ε, επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε μαζί του και να αποφύγουμε ένα κενό στο σύστημα ασφάλεια μετά την αποχώρηση του ΗΠΑ από την Ένωση. Αυτό θα μα συνέφερε όλου. Ευχαριστώ πολύ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Τσινίτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω Αρχικά να ευχαριστήσω τον εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ, την κυρία Ντεμπόλ, για την παρουσίασή της. Όπως τονίσατε, ο ρόλος της Ευρωπόλ έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται όλο ένα και ζωτικότερος στην πρόληψη και την καταπολέμηση των σαβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, της τρομοκρατίας, του κύβερνου εγκλήματος και τόσων άλλων μορφών εγκληματικότητας. Όπως και εσείς οι ίδιοι υπογραμμίσατε, είναι σημαντικότατη συνεργασία με τις εθνικές αρχές για την αναχέτηση ε, και βεβαίως και με τους υπόλοιπους ε, οργανισμούς που εργάζονται στον χώρο του εγκλήματος. Ήθελα να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπόλ στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 ε, ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων. Βάσει της σύστασης του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς σκοπούς για τους οποίους ε, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία η Ευρωπόλ για σκοπούς ε, ανάλυσης των πληροφοριών ή για επιχειρησιακούς. Και τι, ε, πώς εντάσσεται το έγγραφο αυτό το τομέα της διαλειτουργικότητας και της ε, ανάλυσης, της διασυνδεδεμένης ανάλυσης των δεδομένων. Και έπειτα ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα για τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών της Ένωσης. Θέλω να μου πείτε, κατά πόσον έχετε δει τις διάφορες μορφές συνεργασίας που έχει η Ευρωπόλ ε, με την Eurojust και πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Και επιπλέον στο έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021 ε, δεν υπάρχει καμία μνήα της, ας το πω έτσι, μελλοντικής προβλεπόμενης συνεργασίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Ευρωπόλ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, σκέφτεστε τι ε, ανάγκη θα υπάρχει για τέτοιου είδους συνεργασία και τι αντίκτυπο θα έχει και στους πόρους σας εφόσον απαιτηθεί μια τέτοια συνεργασία Ευρωπόλ ε, και Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Και τώρα από τα Εθνικά Κοινοβούλια για την Ιρλανδία. Ο κύριος Οκουίλαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σημειώνουμε κάποια σχετική ανησυχία ότι στο πολιετές της πρόγραμμα Ευρωπόλ όταν αναφέρεται στην ενίσχυση της εταιρικής της σχέσης με τρίτα κράτη, δηλαδή εξωευρωπαϊκά, αναφέρεται στις ΗΠΑ, τις χώρες της Μεσογείου, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Ε, δεδομένου ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει ε, το Μάρτιο του 2019 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό ξεπερνάει το, την πρόπτικη του γράφου προγραμματισμού δεν υπάρχει κάποια μνήμα τη αποχώρηση αυτή στο έγγραφο. Δεν είναι σημαντικό η Ευρωπόλη να έχει μια καλή συνεργασία και με τι αστυνομικέ αρχέ τη Βόρειου Ιρλανδία. γιατί και αυτή η περιοχή θα αποχωρήσει από την Ένωση. Και για την κυρία Ντεμπόλ θα ήθελα να μου πείτε Πώ ε, διαμορφώνονται οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπόλ σε σχέση με την αποχώρηση της Βρετανία και σε σχέση με το σχέδιο προγράμματο για τις ε, νέε ε, τις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων και το προφίλ πρόσληψης των υψηλών αναλυτών και διαχειριστών στην Ευρωπόλ, των μάνατζερ δηλαδή τι θα γίνει με τους διορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν και το πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Ευχαριστούμε κύριο Κούιλαν. Και τώρα κάτω χώρες. Κυρία Ντανμπιόρ. Καλημέρα σας. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ θετικό που βρισκόμαστε εδώ ως μέλη της Βουλής και της Γερουσίας από τις κάτω χώρες και είμαστε όλες γυναίκες, 100%. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Εγώ είμαι από την κάτω Βουλή και δεξιά έχουμε δύο μέλη ε, από τη Γερουσία, η κυρία Βέιζεν και η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ενημέρωση πάντα και πληροφόρηση μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων και για το μέλλον της Ευρωπόλ έχετε φιλοδοξία να γίνετε πιο ε, επιχειρησιακοί από το πολιετές σας πρόγραμμα. Αυτό είναι καλό και πρόσδεκτο, αλλά τι σημαίνει συγκεκριμένα για τα κράτη-μέλη. Τι θα πει full scale delivery των επιχειρησιακών αυτών δυνατοτήτων και επέκταση για την ιδιωτική συνεργασία, για την πολυκλαδική συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό και τι αποτέλεσμα θα έχει. Ε, θα επιθυμούσαμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στα πλαίσια του κράτους δικαίου ε, ε, διερωτώ πόσο είναι επιθυμητή η επέκταση σε τρίτες χώρες που έχουν και κακή φήμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιες συμφωνίες κάνουμε με τις τρίτες χώρες. Τι γίνεται με τις κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων. Πώς διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα και τι γίνεται με τους ε, ταξιδιώτες, τους επιβάτες αεροπλάνων, τα PNR, τη FTT και διάφορες λίστες. Κατά πολέμηση τρομοκρατίας, ε, οι αρμοδιότητές σας ε, είναι εξίσου μεγάλες με τις διοκτικές σας αρμοδιότητες για το έγκλημα και ποια είναι η σχέση των δικών σας αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες των διοκτικών αρχών των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στην Ουγγαρία. Η κυρία Τενάτση, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εκτελεστικοί διευθύντρια, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο εγγράφου ε, προγραμματισμού της Ευρωπόλ εστιάζει στις προκλήσεις της μετανάστευσης και τις απειλές της τρομοκρατίας. Πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα ε, είναι η συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου θεωρούμε ότι είναι καθοριστική σημασία η συνεργασία με την Ευρωπόλ καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με συνεργαζόμενες υπηρεσίες. Είμαστε υπέρ τη ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ε, που χρησιμοποιούν οι άλλες ε, υπηρεσίες και θα θέλαμε να ενισχυθεί η συνεργασία σε λειτουργικά προγράμματα. Το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού της Ευρωπόλ βασίζεται στις προτεραιότητες που ανακοινώθηκαν. Από τις προτεραιότητες που αναφέρονται η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και για την Ουγγαρία. Ε, Εξαιτία της γεωπολιτικής κατάστασης μας, θέσης μας, πρέπει να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα τη διαχείριση των συνόρων του Σέγγεν και να προβλέψουμε την ενδεχόμενη εξέλιξη του εγκλήματος ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ε, διασυνοριακά και η ε, συνεργασία που ε, βασίζονται σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλουμε επίσης ευρωπαϊκή Ευρωπόλ να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός οργανισμός με ε, αποτελεσματική διακυβέρνηση. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης των ε, μέσων και εργαλείων και ταυτόχρονα η συμμετοχή των ε, κρατών μελών να γίνει πιο διαφανής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας σε αυτήν την συνεδρίαση. Ευχαριστώ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Λόρδος Κέρκοπ από την Βρετανική Βουλή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τη νέα Διευθύντρια της Ευρωπόλ υπό την ιδιότητά της. Ασχολήθηκε πάρα πολύ ε, και με τις εκκλήσεις για τη μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι παρόν σήμερα στη συγκεκριμένη ε, δήλωση και συμμετέχω στη διαδικασία. Επίση χαίρομαι πάρα πολύ που κυριολεκτικά πριν από λίγε μέρε το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε το opt-in ε, στο νέο κανονισμό έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών για την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματο χρήματο στην αντίστοιχη τέταρτη οδηγία και εν ώψη τη πέμπτη. Καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσει τη σημασία του Ευρωπαϊκού της Ευρωπόλμα. Ήμουν εισηγητής για το PNR και ε, είναι κρίσιμη ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για το μέλλον της ασφάλειάς μας στην Ευρώπη. Και καθώς πολλαπλασιάζονται οι οργανισμοί με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζεται ε, η Ευρωπόλ και εντός της Ένωσης αλλά και με εξωτερικούς οργανισμούς, ε, ανησυχώ αρκετά Ανεξαρτήτως από την έκβαση της ε, σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου εντός ή εκτός της Ένωσης, θα ήθελα να σχολιάσει η Διευθύντρια ε, στην απάντησή της ε, όλο αυτό το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και τους κανόνες και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις της Ευρωπόλ για τα δεδομένα και την ασφάλεια και πώς όλα αυτά διαβιβάζονται σε μια συνεχιζόμενη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και λοιπόν Ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό με ενισχύει βαθύτατα και καταλαβαίνουμε όλοι πρόεδρε ότι το σημαντικότερο που είναι η επιτυχία της Ευρωπόλου αυτά τα χρόνια ε, συμπεριλαμβάνει την ισχυρή και ε, ενεργή συνεργασία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέντες από τη Γαλλία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η ερώτηση μου είναι πολύ απλή. Πώς η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων η Ευρώπη μπορεί ε, να γίνει ε, η Ευρώπη θα, η Ευρωπόλ θα γίνει μια ε, επιχειρησιακή αστυνομική αρχή στην Ευρώπη. Μπορεί η δράση της Ευρωπόλ να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι. Ευχαριστώ πολύ και για τη συντομία σας, γιατί έχουμε αρκετούς συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Να είστε σύντομοι δυνατόν. Από τις κάτω χώρες και πάλι, η κυρία Μπίζελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η γερουσία των κάτω χωρών θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης, καθώς επίσης και την Ευρωπόλ για τη συνεισφορά της στην καταπολέμηση ε, του εγκλήματος στην Ευρώπη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το πολιετές ε, πρόγραμμα της Ευρωπόλ. Ο δεύτερος στόχος για την επιχειρησιακή υποστήριξη της Ευρώπης λέει ότι η Ευρωπόλ θα πρέπει να δρά υποστηρικτικά στα κράτη-μέλη σε περίπτωση ε, ε, διεκτικών ερευνών. Ποια θα είναι αυτή η υποστήριξη εκτός από την ανταλλαγή προφοριών. Τι διοκτικές αρμοδιότητες θα έχουν οι συνεργάτες της Ευρωπόλ που πηγαίνουν να συμμετέχουν στις έρευνες που κάνουν τα κράτη-μέλη και με ποια εντολή και με ποια πλαίσια και με ποιον τρόπο η δική μας μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου θα τα ελέγχει όλα αυτά και θα τα υποπτεύει. Μπορεί η Ευρωπόλ να μας πει ποιος ήταν ο ρόλος της σε διάφορες αστυνομικές έρευνες. Περιμένω να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι για τη συντομία σα Από τη Βολή των Ελλήνων, ο κύριος Παπαθεοδόρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντεμπόλ, την καινούρια διευθύντρια ε, της ε, ε, Europol, για την ε, πλήρη και πολύ λεπτομερή έκθεσή της σχετικά με το πολιτές πλάνο ήθελα να επικεντρώσω όμως περισσότερο την ε, παρέμβασή μου στις προκλήσεις, στις νέες προκλήσεις που ε, αναδύονται σήμερα, που υπάρχουν σήμερα μεταξύ της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Βεβαίως και δεν βρισκόμαστε πλέον στο 2015. Το 2015 όπου είχαμε μεγάλα ε, προσφυγικά ε, ε, κύματα. Βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που εφαρμόζεται η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και σύμφωνα με αυτή προβλέπεται ή έχει αυτό ως αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλά ελληνικά νησιά ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός προσφύγων. Ένας πληθυσμός που σήμερα μόνο σε πέντε νησιά φτάνει τους 15-18 χιλιάδες πρόσφυγες αυτή η σχέση με την προσπάθεια της europol αλλά και την προσπάθεια πολλών ευρωπαϊκών ε, μηχανισμών να αντιμετωπίσουν ε, την προσφυγική κρίση θεωρώ ότι θα φέρει μεγαλύτερη ανασφάλεια και μάλιστα σε μια περίοδο όπου λόγω της προεκλογικής περίοδου των ε, ευρωεκλογών θα συζητηθεί πολύ το θέμα της ασφάλειας και της σχέσης που έχει με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής ποια είναι τα μέσα τα επιπλέον μέσα που η ε, europol μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμερα για να αντιμετωπίσει κινδύνους ανασφάλειας οι οποίες έχουν να κάνουν με την ε, προσφυγική κρίση και αν νομίζει αν έχουμε συνειδητοποιήσει πως τέτοιου είδους ε, διαχείριση στο προσφυγικό τελικά θα φτάσει σε μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση μεγάλων ομάδων του προσφυγικού ε, πληθυσμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Ισπανία ο κύριος Τολετάνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ. Σύντομα κάποια σχόλια και μερικές ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπόλ, όπως ε, γνωρίζουμε και όπως ακούσαμε. Κατά πολέμηση τρομοκρατίας, κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ηλεκτρονικό έγκλημα, οι διάφορε μαφίες ε, των διακινητών, μεταναστών. Όλα αυτά κάνουν την ισπανική αντιπροσωπεία να ανησυχεί για αυτά που ακούσαμε σχετικά με τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχετε ως οργανισμός για την ε, πληροφόρηση, το συντονισμό και την ε, συνεργασία και τη συμμετοχή με τις εθνικές αστυνομίες για την καταπολέμηση αυτών των τόσο σοβαρών εγκλημάτων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πού οφείλεται αυτή η υποχρηματοδότηση. Οφείλεται εν μέρη στο Brexit, στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου και πώς μπορεί να λυθεί οικονομικά αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, γιατί μας ανησυχεί ότι μπορεί να έχει ανετικές επιπτώσεις για την ασφάλεια της χώρας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές στα μάτια των πολιτών ε, υποφέρει από άγνοια των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας της. Και για να μπορέσει να αυξηθεί το κύρος της και η εκτίμηση ε, στα μάτια των πολιτών βοηθάει το να γνωρίζουν οι πολίτες αυτούς τους οργανισμούς και μεταξύ αυτών είναι η Ευρωπόλ. Καλό είναι να γνωρίζουν οι πολίτες τι κάνουν οι οργανισμοί αυτοί και πώς η Ευρωπόλ βοηθάει στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών μας. Αυτό σίγουρα ε, θα επέτρεπε ένα καλύτερο συντονισμό και αύξηση της πίεσης για να αυξηθούν και τα κονδύλια σας. Και μια τελευταία ερώτηση προσωπική. Πώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κατά την απόψή μου η κρίση που γνωρίσαμε πρόσφατα με τα ευρωεντάλματα σύλληψης. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Η κυρία Καραμαλή από τη Γαλλία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι όλες οι παρεμβάσεις των συναδέλφων δείχνουν την ανησυχία που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ε, λειτουργία και τις δυνατότητες συνεργασίας. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην ε, Ευρωπόλ και τις άλλες υπηρεσίες ε, θα υλοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει επικάλυψη ανάμεσα στην Ευρωπόλ και την Frontex που θεωρεί επίσης ε, την καταπολέμηση της τρεμοκρατίας και της διακίνησης όπλων προτεραιότητα παρόλο που η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ε, είναι η βασική της αποστολή καθώς και σε ό,τι αφορά την κατανομή των ρόλων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Επίσης κυρία Διευθύντρια, ε, η εμπειρία που αποκτήσατε ε, στα hot spot ε, ίσως ε, μπορεί να χρησιμεύσει για την ανάπτυξη αυτών των νέων κέντρων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Θα θέλαμε λοιπόν αυτό το θέμα να το κοιτάξουμε πώς θα αποφευχθεί η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και πώς θα καλυφθούν οικονομικά ε, αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πριν δώσουμε ε, το λόγο στην κυρία Ντεμπόλ, τελευταίος ο κύριος Έγγελ από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ντεμπόλ για την παρουσίασή τη και για όσα πέτυχε στο πεντάμινο ε, άσκηση των καθηκόντων τη. Θα πρέπει να τη πω ότι και σε επίπεδο συμβουλίου βλέπουμε ότι όλοι ζητάνε περισσότερα ε, και με, πάντοτε με λιγότερους πόρους. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπόλ. Αλλά σε σχέση με, το, ε, με την εικόνα που διαμορφώνεται για τους πόρους σας μελλοντικά, εγώ είμαι υπέρ της υπηρεσίας αυτής της Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε πολλούς οργανισμούς και υπηρεσιέ της Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε οι υπάλληλοι να αντικαθίστανται από ε, προσωρινούς υπαλλήλους ή συμβασιούχους. Στην Ευρωπόλ Ποια είναι η έκταση αυτού του φαινομένου, γνωρίζοντα ότι πολλοί από αυτού που εργάζονται για την Ευρωπόλη είναι αποσπασμένοι από τα κράτη-μέλη αλλά χρειαζόμαστε ε, υπαλλήλου με πραγματικά ισχυρή κινητοποίηση και διάθεση να δουλέψουν για την Ευρωπόλη και να αφοσιωθούν στο σκοπό τη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τι τόσο εύστοχε ερωτήσει σα και τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα με ιδιαίτερη χαρά θα δώσω το λόγο στην εκτελεστική διευθύντρια. Έτσι για να έχουμε μια ιδέα, στις 5 θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της συζήτησης, οπότε ξέρω ότι δεν θα καταφέρετε να απαντήσετε σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά τα περισσότερα από τα θέματα αυτά είναι μεγάλης ε, εμβέλειας, οπότε είναι και σε εξέλιξη και απαντήστε όπως νομίζετε εσείς, Κάθριν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε ε, την υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεκινώντας με το μεταναστευτικό. Η μετανάστευση, η Ευρωπόλ έχει ένα ειδικό κέντρο για τη διαχείριση της ε, μετανάστευσης ε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 90 έρευνες που αφορούν διακινητές μεταναστών σε υψηλό επίπεδο. Αυτές είναι οι δυνατότητες μας αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τις δευτερεύουσες ε, κινήσεις, ε, το εξετάζουμε αυτό το θέμα. Αυξάνονται τα, οι δυσκολίες Παραμένουμε σε επαγρύπνηση. Μια ενίσχυση της προσέγγισης για τη, της επιχειρησιακής μας δράσης σε ό,τι αφορά τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών είναι όντως απαραίτητη. Θέλουμε οι δράσεις μας να είναι αποτελεσματικές. Μία παρουσίαση ε, με τα δέκα βασικά θέματα θα γίνει στο Συμβούλιο. Θα υπογραμμίσω τρία από αυτά θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μιας ε, task force για τη διαχείριση της μετανάστευσης ε, στα πλαίσια συνεργασίας της ε, Ευρωπόλ και των κρατών μελών. Θα το κάνουμε, το κάνουμε ήδη στο τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχουμε αποτελέσματα γιατί οι ερευνητές μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συζητήσουν. Δεύτερον, θέλουμε να επικεντρωθούμε στα κέρδη των διακινητών. Πρέπει να εστιάσουμε περαιτέρω σε αυτό το θέμα πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες σε διάφορα κράτη-μέλη ε, με μεγαλύτερη συχνότητα προκειμένου να εντοπιστούν οι διακινητές και ε, να δεσμεύσουμε ε, τα περιουσιακά του στοιχεία. Θα υποστηρίξει αυτή τη δράση η Ευρωπόλ. Η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της δράσης των διακινητών πριν φτάσουν οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών ε, με τις τρίτες ε, χώρες. Ε, πρόκειται για θέμα πρωταρχικής σημασίας, άμα θέλουμε να είναι αποτελεσματική η δράση μας σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τη διαφθορά, το γεγονός ότι η διαφθορά δεν αναφέρεται τον πολιετή προγραμματισμό μας. Πράγματι, ε, η διαφθορά ε, σχετίζεται με όλα τα ε, τις μορφές εγκληματικής δραστηριότητας Κάποιες έρευνες σε ορισμένες ε, χώρες ε, είχαν να κάνουν με αυτό το θέμα τους τελευταίους μήνες. Πρέπει να ορίσουμε ακριβώς την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στους ε, αστυνομικούς η Ευρωπόλη σε ό,τι αφορά την ένταξη της διαφθοράς στο έγγραφο προγραμματισμού και στο πρόγραμμα εργασιών του 2019 Ήδη έχουν προβλεφθεί κάποιες ε, εργασίες. Η Ευρωπόλ θα ε, υποστηρίξει την καταπολέμηση της διαφοράς στα κράτη-μέλη και θα ενισχύσει τη συνεργασία της Ευρωπόλ με τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ε, σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία. Έχει υπογραμμαστεί αυτό το θέμα από τον εκπρόσωπο του ε, Κυπριακού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για θέμα προστιθέμενης, ε, που θα προσφέρει προστιθέμενη αξία η συνεργασία. Η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπόλη και την ε, Τουρκία βασίζεται σε στρατηγική συμφωνία που ξεκίνησε το 2014. Αποκλείεται όμως η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Διευκολύνεται η συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς και έχουμε έναν ε, αξιωματικό σύνδεσμο από την Τουρκία στα γραφεία μας. Ξεκίνησε τη θητεία του το 2016 2016, αλλά η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων δεν είναι δυνατή. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική συνεργασία, πρόκειται για αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με τη Τουρκία για την ανταλλαγή ε, προσωπικών δεδομένων με τη Τουρκία. Η Τουρκία έχει ενταχθεί στις χώρες προτεραιότητες, ε, όπως και το αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο το ή ε, είχε ε, επιτυχή αποτελέσματα, πολύ θετικά. Ξεκίνησε το 2015 και μέχρι σήμερα ε, έχει οδηγήσει 64.000 αναφορές την τελευταία εβδομάδα ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, ανακοίνωσε τη δημοσίευση ενός σχεδίου κανονισμού για την καταπολέμηση της ε, ε, ε, ε ριζοσπαστικοποίησης στο διαδικτύο θα εξετάσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί η σχετική ε, πλατφόρμα, όπως και να ε, θα χρειαστούν ε, και οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι. Έχει επικοινωνήσει μαζί μας η Επιτροπή σε ό,τι αφορά πριν την παρουσίαση αυτής της πρότασης και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ λίγος ο διαθέσιμος ε, χρόνος. Είναι ε, πολύ σημαντική το θέμα αυτό για την αντιμετώπιση της ριζοσπατιστικοποίησης. Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές ότι κάποιες φορές θα υπάρχει επικάλυψη στη δράση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εργαστούμε πάνω σε κοινέ στρατηγικές και αξιολογήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουν ταυτόχρονα τα διοικητικά συμβούλια της Frontex και της Ευρωπόλ. Θα εξετάσουμε τις αρμοδιότητες των δύο υπηρεσιών και θα εξετάσουμε τις δυνατότητες ε, συνεργασίας. Είμαι πεπισμένη ότι σε υψηλό επίπεδο η συνεδρίαση θα είναι εξαιρετική με τη Frontex και εδώ ότι θα βρεθούν λύσεις. Οι δύο υπηρεσίες έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Η Ευρωπόλ είναι κόμβος ανταλλαγής ή ε, πληροφοριών σε ποινικέ ε, έρευνες. Η Frontex ε, έχει ως αποστολή την προστασία των συνόρων μας. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες είναι πρωταρχική σημασία και θα ληφθεί υπόψη αυτό στο μέλλον. The financial crime. Η υπηρεσία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματο ε, είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα. Και το βλέπουν διαφορετικά οι διάφοροι αρχηγοί αστυνομιών, αλλά θέλουν να επενδύσουμε στην καταπολέμηση αυτού του είδους εγκλήματο και να βοηθήσουμε την εκπαίδευση των αστυνομικών για να μπορούν να κάνουν σχετικέ έρευνε. Στο επίπεδο τη Ευρωπόλη είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα Γι' αυτό θα αξιοποιήσουμε όλη την ε, εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπόλ αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με οκτώ ε, υπηρεσίες, εθνικές υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος και έχουμε δει πολύ καλά αποτελέσματα. Η Ευρωπόλ ακολουθεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, της, Επιτροπή, της Επιτροπής, για τους όρους και τις προποθέσει των πληροφοριών σε σχέση με τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και έτσι ε, έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα από τις εθνικές υπηρεσίες μέσω της δικής μας ε, κεντρικής υπηρεσίας. Πρέπει πάντοτε να περάσουμε όμως ε, από την Ευρωπόλη στην Εθνική Υπηρεσία, την ομόλογη, και πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα είναι ένα περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Όπως είπα, είναι προτεραιότητα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον προπολογισμό το 2019 ήδη υπογράμμισε και ο Πρόεδρος και πολλοί από τους ομιλητές σε αυτό το γύρο συζήτησης ότι το σχέδιο προπολογισμού για το 2019 προβλέπει κονδύλια ε, για την Ευρωπόλ 120,9 εκατομμύρια με 5 μόνο επιπλέον θέσεις. Δεν λαμβάνει υπόψη Πολλέ από τις πρωτοβουλίε που πρέπει να αναπτύξουμε, πολλές από τις πρωτοβουλίε που μας έχουν ζητηθεί να αναπτύξουμε. Ε, η πρόταση λοιπόν του προπολογισμού έχει μείωση μάλιστα 8,2 εκατομμύρια σε σχέση με τον προπολογισμό του 2018. Η περικοπή αυτή φτάνει τα 21 εκατομμύρια εάν τη συγκρίνουμε με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ. Οπότε, εάν ε, η πρόταση του προπολογισμού ε, που έχουμε κάνει εμεί δεν γίνει δεκτή, το πρόβλημα είναι ότι η αξιωματικοί που έχουμε αποστείλει στα hot spot, που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων, ε, δεν θα μπορεί να ε, προχωρήσει. Ε, επίση, η πλατφόρμα για την αποκρυπτογράφηση πληροφοριών που έπρεπε να ξεκινήσει το 2018 και είναι σημαντική για την καταπολέμηση του κυβερνού δεν θα προχωρήσει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε ευρωπαϊκή κλίμακα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών. Και επίση για την ενίσχυση των συστημάτων μα πληροφορική. Δεν θα έχουμε την απαραίτητη πρόοδο έχουμε ακόμη δυσκολίες στην υποστήριξη της δουλειάς των κρατών μελών στις ειδικές ομάδες ε, δράσης. Μια από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της ομάδας Atlas, το δίκτυο Atlas όπως έχει ονομαστεί, μας είχε μάλιστα καλέσει η Προεδρία να τις ενισχύσουμε για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Απαιτούνται πόροι και γι' αυτό. Εάν Θέλουμε ε, επίσης το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο να απομακρύνεται, να διαγράφεται αμέσως, πάλι χρειάζονται ε, έλεγχοι που να μπορούν να γίνονται γρήγορα. Ακόμη και για τους ελέγχους στα hot spot ε, χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας του σκοτεινού δικτύου επίσης είναι κάτι που απαιτεί πόρους, απαιτεί δουλειά και χρήμα. Όπως είπα, τα συστήματα πληροφορική μα τα τελευταία χρόνια δεν έχουν προχωρήσει όπω θέλαμε, δεν έχουμε επενδύσει ακόμα, διότι όποτε χρειαζόμασταν επιπλέον χρήματα, τα κόβαμε από το κονδύλι για, το, για τους υπολογιστέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποστήριξη, γιατί τα νέα κρατημέλη ζητούν την υποστήριξη των παλιών για να μπορέσουν να αναπτύξουν τι δικέ του δυνατότητε στην αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών, την διασύνδεση και την ανάλυση των πληροφοριών. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά και να μπορέσουμε να τα συντονίσουμε, θέλουμε να έχουμε πόρου για τον Brexit. Πολλοί από τον χώρο των ιδιοκτικών αρχών ανησυχούν Ω προς τον Brexit. Έχουμε ήδη κάνει κάποια βήματα για να προβλέψουμε τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit και έχουμε θέσει και επιμέρου, επιμέρους ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όμως τον απόϊχο του Brexit, ε, τους τριγμούς θα προκαλέσει και όλα τα ζητήματα θα προκύψουν, διότι η λύση είναι απαραίτητη. Ε, η λύση είναι απαραίτητη, μάλλον στην εξέβρεση λύση είναι απαραίτητη η συμμετοχή τη Ευρωπόλη, προκειμένου να διατηρήσουμε το ε, σκηνικό ασφάλεια που γνωρίζουμε. Όλα τα πιθανά σενάρια σε σχέση με τον Brexit βρίσκονται επιτάπητο και συζητώνται. Θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συζητάμε και με του αρχηγού αστυνομιών για τι διαφορετικέ ε, προοπτικέ που μπορούν να διαμορφωθούν λόγω του Brexit. Η ερώτηση για την ολοκληρωμένη την κοινή διαχείριση των δεδομένων. Ο ρόλος της Ευρωπόλ εδώ ποιος είναι. Είναι ο σκοπός της ανταλλαγής πληροφοριών. Πρέπει να καθορίζει το σκοπό. Και εδώ έχουμε τέσσερις διαστρωματώσεις. Πρώτα απ' όλα διασταυρούμενο έλεγχο των δεδομένων. Δεύτερον, στρατηγική και θεματική ανάλυση των δεδομένων. Τρίτον, επιχειρησιακή ανάλυση. Και τέταρτον, διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. Άρα η βάση δεδομένων που έχει αναπτύξει η Ευρωπόλ ήταν ένα τέτοιο σύστημα που ελάμβανε υπόψη αυτές τις τέσσερις διαστρωματώσεις. Ε, τώρα θα πρέπει το σύστημα αυτό να ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό για τον οποίο ζητά κάποιος τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η προστασία των δεδομένων είναι επίσης σημαντική και η προσπάθεια που κάνουμε τώρα έχει να κάνει με του όρου που προέκυψαν από την προστασία δεδομένων. Σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ε, οι κανόνε που έχουν προκύψει είναι πολύ αυστηροί και έχουμε πολλού επόπτε και επιθεωρητέ, φορεί και σώματα που εποπτεύουν. Ε, ταυτόχρονα στην Ευρωπόλη έχουμε και ανεξάρτητο ε, επιθεωρητή δεδομένων, ε, διαχείριση δεδομένων τον έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθημερινώς διατρέχει τα συστήματά μας για να δει εάν συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες ή όχι. Εάν όχι, λογοδοτούμε. Εξωτερικώς έχουμε τον Ευρωπαϊκό Επόπτη ε, Προστασίας Δεδομένων, EDPS, και έχουμε διαμορφώσει μια ισχυρή σχέση μαζί τους. Έχουμε και τις εθνικές αρχές ε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, καθώς και ένα συμβούλιο συνεργασίας. Η Ευρωπόλ έχει λοιπόν θέσει κανόνες και του στηρεί για την ε, παροχή και την διαχείριση των δεδομένων, για την επεξεργασία τους και για την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα ε, τα παραλαμβάνουν μόνο οι παραλήπτες που έχουν ε, νομικός και νομίμως το δικαίωμα να τα παραλαμβάνουν και βρίσκονται μόνο στα χέρια των κρατών μελών, των υπευθύνων τους. Υπεύθυνο δε είναι ο Μάλλον κάτοχος των δεδομένων είναι αυτός που τα αποστέλει. Αυτός είναι νομικά υπεύθυνο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι στην ουσία οι κάτοχοι των δεδομένων, οι υπεύθυνοι. Η πρόσβαση των δεδομένων διευθετείται από τις εσωτερικές κατευθυντήριε γραμμέ επεξεργασία δεδομένων τη Ευρωπόλ και οι μόνοι που μπορούν να τα δουν είναι όσοι έχουν εξειδίκευση στο χώρο αυτό ή έχουν λάβει ειδική άδεια ή έχουν ε, ήδη εργαστεί στο χώρο αυτό. Εάν το επιθυμείτε μπορούμε να σας δώσουμε και γραπτές λεπτομερείς απαντήσεις για το ερώτημα αυτό. Ε, νομίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ε, και εγώ αυτό νομίζω. Ναι, βέβαια κάποιες ερωτήσεις απαιτούσαν λεπτομερέστερες απαντήσεις ίσως, αλλά εάν θεωρείτε ότι είναι κάτι σημαντικό που σας διέφυγε και δεν προλάβατε, στα πλαίσια της λογικής, απαντήστε. Ε, η εκτελεστική διευθυντήρια προφανώς θέλει απαντήσεις στις ερωτήσεις όλων σας, οπότε αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ, αλλά Α πούμε για το θέμα του Brexit. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπόλ έχει κάνει ό,τι μπορεί, έχει προετοιμαστεί και σε σχέση με όσα έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι δυσχερή στι διαπραγματεύσει και για το πώ θα διαμορφωθεί η συνεργασία τη ασφάλεια. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά η Ευρωπόλ μέχρι να υπάρξουν κάποιες πολιτικές ε, αποφάσεις. Οπότε είναι πολλά τα κανθόδια ερωτήματα εδώ για την Ευρωπόλ, αλλά Παρακαλώ συνάδελφοι, εάν έχετε ερωτήσεις ε, προχωρήστε, αλλά όλες οι ερωτήσεις σας ήταν εύστοχες. Στα δύο λεπτά που μας μένουν λοιπόν, θέλετε κάτι να προσθέσετε κυρία Ντεμπόλ, εν είδη συμπεράσματος. Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλες τις ερωτήσεις. Ε, πραγματικά ε, έρχονται και ως συνέχεια των συζητήσεων που είχαμε τους υπουργού της Διαφορε Συνδρία του Συμβουλίου και με τους υπευθύνου των ε, εθνικών αρχών και των αρχηγών αστυνομιών και τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε συζητήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους από τα κράτη-μέλη και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτα τα κράτη. Είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του συστήματος ανταλλαγής. Πάντως πραγματικά σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον σας και για το γεγονός ότι ε, σας απασχολεί η επιχειρησιακή στήριξη που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπόλ στα διάφορα κατημέλη και αν μπορώ να απαντήσω ερωτήσει εφόσον έχετε ακόμη απορίε, γραπτός θα το κάνω. Είμαι στη διάθεσή σα να απαντήσω οτιδήποτε θέλετε όταν επισκεφτείτε την Ευρωπόλ. Ελάτε και θα σα τα πω όλα λεπτομέρω. Θα σα πω και άλλα σε σχέση με αυτά που είπα σήμερα εδώ. Ε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν και ελπίζω να σα δω σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ την εκτελεστική διευθύντρια αν έχετε και άλλες ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν έτσι εκ παραδρομής ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, μην διστάσετε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στη γραμματεία ή στην εκτελεστική διευθύντρια απευθεία. Για τα Brexit, αυτά που έλεγα και για την ασφάλεια, το ειδικό θέμα της Europol είναι αυτό που έχει να κάνει με το κατά πόσο θα έχει πρόσβαση το Βασίλειο στη βάση δεδομένων ή μπορεί να είναι μέλος της Ευρωπόλ. Είναι γνωστά τα ζητήματα, αλλά οι διαπραγματεύσεις ε, για τα θέματα αυτά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί προφανώς, ούτε ε, όμως υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη θέση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι πρέπει να αναμένει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επιχειρησιακά είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία Ευρωπόλ αν δεν υπάρχει πρόοδος. Είναι μέγα ζήτημα όμως για τα κράτη-μέλη, όπως είπατε και πολλοί από εσά. Ωραία. Και τώρα θα περάσουμε ε, στο τελευταίο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης. Έχουμε ε, και άλλους ομιλητές και ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ Μάρτιο με Σεπτέμβριο 2018. Θα ακούσουμε τον κύριο Πρίτ Πάκνα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μια αναφορά από τον κύριο ε, Τσβέταν Τσβετάνοφ. Ελάτε παρακαλώ και οι δύο εδώ στο Προεδρείο. Να σας ε, κάνω μια εισαγωγή στο σημείο αυτό και πάλι είναι μέρος της επίσημης διαδικασίας βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού της Ευρωπόλ. Ο κ. Τσφετάνοφ πήρε μέρο στην 107η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Σόφια στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2018 υπό την ιδιότητά του. Γι' αυτό θα συντονίσει και αυτό το μέρο τη συνεδρίαση τη ΜΟΚΕ. Και βέβαια του αρθρό 51 του κανονισμού τη Ευρωπόλ, ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπόλ έχει προσκληθεί για ανταλλαγή απόψεων. Η συζήτηση αυτή και πάλι θα ακολουθήσει το γνωστό ε, σύστημα. Θα δώσουμε το λόγο εναλλάξ. Θα δίνουμε μάλλον το λόγο εναλλάξ σε δύο μέλη εθνικών κοινοβουλίων και σε έναν ευρωβουλευτή. Βεβαίω, αν είναι περισσότεροι οι εθνικοί βουλευτέ, θα είναι μακρύτερο ο κατάλογο των αγορητών. Λοιπόν, πρώτα δίνουμε το λόγο στον κύριο Πριτ Πάρκνα, πρόεδρο του ε, Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπόλ, για 10 λεπτά το πολύ. Κύριε Πριτ Πάρκνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα εξ αρχή να πω ότι 10 λεπτά για να σας μιλήσω για όλο το έργο της Ευρωπόλ το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Νομίζω ότι θα υπερβώ το χρόνο με την αδειά σα φυσικά. Αξιότυπα μέλη τη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα... Είναι ήδη τρίτη φορά που ε, παρεμβαίνω ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ. Υπάρχει νομίζω ένα μικρό πρόβλημα με την ε, διερμηνία. Μπορείτε να μιλήσετε όλες τις γλώσσες εκτός από τα Ολλανδικά. Όλα εντάξει. Ναι. Μπορείτε να συνεχίσετε. Παρακαλώ, συγγνώμη για την ε, που σας διάκοψα. Αυτή η συνεδρίαση της ε, ΜΟΚΕ είναι σίγουρα η τελευταία στην οποία συμμετέχω ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία μου ε, λύγει το Δεκέμβριο και ένας νέος πρόεδρος ε, θα εκλεγεί από την Τριάδα Προεδρίων και θα εκλεγεί και νέος ε, ε αντιπρόεδρος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω, όπως και προηγουμένως, το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η ΜΟΚΕ είναι βασικός εταίρος για τη διασφάλιση του έργου της Ευρωπόλ. Ρόλοι μας είναι πολύ συγκεκριμένοι σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη ε, μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στο τομέα της ασφάλειας και ε, προσδοκούμε η Ευρωπόλη να στηρίξει ακόμα περισσότερο τη δράση των διοκτικών αρχών και να ενισχύσει τη συνεργασία της. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια επισκόπηση των τελευταίων δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη συνεργασία με τη ΜΟΚΕ και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίας στις 3 και 4 Μαΐου του 2018 στη Βουλγαρία, μιας και η Βουλγαρία είχε την Προεδρία, συνεδρίας στη Σόφια. Εξετάσαμε διάφορα θέματα διακυβέρνησης, διοικητικά, επιχειρησιακά ζητήματα και συγκεκριμένα το θέμα της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Και αυτό θα ήθελα να αναφέρω τώρα, σε ό,τι αφορά την διοίκηση και τη διακυβέρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα πολιτική προστασίας της ε, αξιοπρέπειας των ανθρώπων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την σεξουαλική κακοποίηση. Στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπόλ ε, δημιουργήσαμε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο και υποχρεώσει ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ε, ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2017 είχαμε θετικά αποτελέσματα, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τους οικονομικούς πόρους και τη διοίκηση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε με βάση μια γραπτή διαδικασία τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ε, για την ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που δίνουν ε, τα κράτη-μέλη στην Ευρωπόλ. Αυτή η έκθεση αποτελεί μια καινοτομία. Βασίζεται στο άρθρο 7, παράγραφο 11 του κανονισμού της Ευρωπόλ. Αυτή η πρώτη έκθεση αφορά το 2018, θα δημοσιευτεί το 2019. Είμαι πεπισμένος ότι η παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων σε αυτή την ετήσια έκθεση θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην Ευρωπόλη και τα κράτη-μέλη. Η έκθεση αυτή θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και σε όλες τις αρχές που προβλέπονται ε, στο κανονισμό, καθώς και στην ε, ΜΟΚΕ. Και τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω σύντομα για τις ε, την εξέλιξη των δράσεων της Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το, τη συνεργασία, τα κριτήρια συνεργασία με την Αλβανία, τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη και τη Σερβία σε ό,τι αφορά τη τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων πρόκειται για μια καινοτομία που θα βελτιώσει τη συνεργασία με αυτέ τι χώρες Κυρίω ό,τι αφορά τους αξιωματικού συνδέσμού, θα εργαστούμε πάνω στις ε, σχετικές αξιολογήσεις μέχρι το 2019 Επίση, η συνεργασία με τι χώρε των Δυτικών Βαλτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για θέμα πρωταρχικής σημασίας και αυτές τις χώρες, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία ε, απασχολούν τις αρχές. Έχουμε επίσης μια έκθεση σχετικά με τις τάσεις ε, της ε, τρομοκρασίας ε, που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπόλ. Πιστεύω ότι η πρόοδος μέχρι τώρα η πρόοδος ήταν πολύ θετική και έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε αυτές τις χώρες στην δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να συνεχίσουμε έναν διάλογο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού της Ευρωπόλ έχουμε μια εξωτερική στρατηγική που περιλαμβάνει τις προτεραιότητες για το 2017-2020 λάβαμε μία απόφαση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπόλ και την, αρχές, τις διεκτικές αρχές του Ισραήλ. Υπογράψαμε στις 17 Ιουλίου μία συμφωνία πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι η εμβάνθηση των τομέων συνεργασίας σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις εκθέσεις ενημέρωσης, τις αξιολογήσεις, τις διαδικασίες έρευνας, τις τεχνικές πληροφορίες καθώς και τις ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο. Ε, τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, τη διαβούλευση και την υποστήριξη ποινικών ερευνών. Πρόκειται για τους τομείς που εξετάσαμε σε ό,τι αφορά το προϋπολογισμό. Πρώτα όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πίτερ Βίντιγκερ, τον εκπρόσωπο της Αυστρίας και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και για το έργο τους σε αυτό το τομέα. Ε, στη συνεδρίαση του Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις του ε, προϋπολογισμού της Ευρωπόλη για το 2018. Έχουμε πολύ ε, σημαντικές δράσεις που προβλέπονται το επερχόμενο διάστημα. Έχουμε υλοποιήσει Έχουμε τοποθετήσει αξιωματικούς ε, στις ε, δύσκολες ζώνες της ε, Μεσογείου και έχουμε ενισχύσει τις ικανότητες αποκρυπτογράφησης της Ευρωπόλ. Ε, μας στήριξε ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης και όπως είπε η κυρία Ντεμπόλ οι οικονομικές προοπτικές για το 2019 μας απασχολούν. Επιστήσαμε την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Αυστριακής Προεδρίας και του Επιτρόπου για τα ε, θέματα εσωτερικής πολιτικής και μετανάστευσης ε, ε, σε ό,τι αφορά την τη δράση και τη σημασία της δράσης της Ευρωπόλης ε, σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τη διασύνδεση των ε, συστημάτων πληροφοριών και την ε, συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας καθώς και τη συνεργασία με τους παρόχους ίντερνετ. Έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 21 εκατομμύρια περικοπές και κατάργηση 38 θέσεων σε αυτό το σχέδιο ε, προβλέπονται. Γι' αυτό σας ζητώ σήμερα την υποστήριξή σας θα είναι καθοριστική σημασία ε, η υπεράσπιση του προπολισμού του, της Ευρωπόλ προκειμένου η υπηρεσία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή δράση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήθελα επίσης ε, να εξετάσω, να εξετάσω το θέμα της ε, συνεργασίας ανάμεσα στη ΜΟΚΕ και, και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινοβουλίου ε, ε, ε, συμμετείχε ο κύριος Τσβετανόφ, τον οποίο ευχαριστώ για την υποστήριξή του. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του κυρίου Τσβετανόφ και θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα τα θέματα που αναφέρθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση του Δυτικού Συμβουλίου καθώς και ε, στα πλαίσια των προπαρασκευτικών εργασιών για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όχι μόνο πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία αλλά χρειάζονται και ε, ε, χρειάζεται και ε, ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει πραγματικά να τηρήσουμε τον κανονισμό της Ευρωπόλ. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να λειτουργήσει ως κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπόλ να, να υλοποιηθεί η εποπτεία του οργανισμού, να προβληθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και, να, ε, και οι ε, ε, απαντήσεις που επιτρέπουν την λειτουργία, την αποτελεσματική λειτουργία των αρχών των κρατών μελών. Και αυτό για να ε, υλοποιηθεί η εποπτεία της δράσης των Ευρωπόλ με διαφανή τρόπο, ενισχύοντας ε, την δημοκρατική νομιμότητα καθώς και τη λογοδοσία απέναντι στους Ευρωπαίους ε, πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο συνειδητοποιούμε ότι η ΜΟΚΕ είναι πρωταρχικής σημασίας μιας και έχει την αποστολή να αποκτήσει πληροφορίες. Μόνο έτσι μπορεί να υλοποιηθεί ο έλεγχος ε, σε όλη την Ευρώπη και αυτό διευκρινίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπόλ, συγκεκριμένα η ΜΟΚΕ. Στις συνεδριάσεις με την Ευρωπόλ πρέπει να έχει όλες τις πληροφορίες ε, για τις ε, δράσεις του οργανισμού και να επικοινωνεί με τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπόλη. Γι' αυτό εκτιμώ τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να σας ε, ενημερώσω προκειμένου να μπορέσετε να ελέγξετε τη δράση μας. Έχω τη τιμή να σας παρουσιάσω και να σας πω ότι τα τελευταία έγγραφα, όπως ε, το έγγραφο προγραμματισμού 2019-2017, η ετήσια έκθεση πεπραγμένου του 2017, μας επιτρέπει να συμμορφωθούμε και να λειτουργήσουμε με βάση το πολιετές πρόγραμμα 2019-2021. Συνεχίζεται η ε, μεταφορά πληροφοριών στην ε, ΜΟΚΕ και ε, αναμένουμε ανυπόμονα την, τις παρατηρήσεις σας σχετικά με αυτά τα θέματα. Η εκπροσώπηση της ΜΟΚΕ στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας πω ότι βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 4 του κανονισμού της Ευρωπόλ, μπορεί να ε, κληθεί να συμμετάσχει ε, κάποιος ε, παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου όμως ως ό,τι αφορά τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στις 4 Μαΐου ο κύριος Τσετάνοφ παρουσίασε την ανάγκη ε, αυστηρής ερμηνείας του άρθρου 14 σε ό,τι αφορά ε, το έργο ελέγχου του, της ε, ΜΟ και προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με το κανονισμό της Ευρωπόλ. Σας μίλησα για το άρθρο 14 το οποίο αφήνει κάποιο περιθώριο στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ε, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις του παρατηρητές είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας. Ακούσαμε τις απόψεις ε, της ΜΟΚΕ και στη συνέχεια εργαστήκαμε προκειμένου να διατυπώσουμε μία ε, τελική ε, πρόταση εν ώψη της συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στι 3 και 4 Οκτωβρίου του 2018. Ε, ξεκίνησε μία γραπτή διαβούλευση με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ε, που θα αφορά τη συμμετοχή ενός ε, μέλους της ΜΟΚΕ Ε, πρόκειται για τη δυνατότητα μόνιμης εκπροσώπησης ε, της ΜΟΚΕ στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω μια οριστική απόφαση γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαβούλευσης. Στη συνεδρίαση στις 3 Οκτωβρίου θα ληφθεί σχετική απόφαση και θα ε, ενημερώσω σχετικά την ε, ΜΟΚΕ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα τις δυνατότητες που δίνει το άρθρο 14 του κανονισμού. Για παράδειγμα, μπορούμε να ε, προβλέψουμε το γεγονός ότι η Ευρωπόλ θα διζητήσει γνωμοδότηση από τη ΜΟΚΕ στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για το πολιετές προγραμματισμό της Ευρωπόλ. Πρόκειται για σημαντικό θέμα και συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τον κύριο Τσφετανόφ. Πρέπει να βρεθεί ένα κοινό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ε, γίνει διαβούλευση με το ε, τιμό και σχετικά με το πολιετές ε, πρόγραμμα της Ευρωπόλ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δημιουργίας μιας πλατφόρμας, <clears throat> είναι κάτι θετικό. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να βρούμε μια καλή ε, φόρμουλα έτσι ώστε η ΜΟΚΕ να συμμετέχει ε, σε αυτές ε, τις συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις μας χρειάζονται την παρουσία της ΜΟΚΕ για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι θα πιάνει και τόπο η δουλειά αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπιστευτικό ή απόρριτο χαρακτήρα των συνεδριάσεων μας, ε, αυτά αφορούν θέματα που δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί ε, και πληροφορίες που είναι για εσωτερική χρήση και όχι για δημοσίευση. Επιπλέον, τα έγγραφά μας μπορεί να αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες, διαβαθμισμένες σημεί για επιχειρήσεις που τρέχουν. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται και να μην δημοσιεύονται ή να μην κοινοποιούνται. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση ε, που ε, θα συνάδει και θα ε, προσαρμόζεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπόλ. Είμαι πεπισμένο ότι θα βρούμε μια λύση για όλα τα πρακτικά ζητήματα πάντα σε συνεργασία ε, μεταξύ μας. Ε, τα μέλη της ε, δική σα ομάδας, της ΜΟΚΕ, έκαναν σχόλια σχετικά με τις γλώσσες που χρησιμοποιούμε στις συνεδριάσεις μας. Ξέρετε ότι για το γλωσσικό είναι αρκετά περιορισμένοι οι πόροι μας και θα πρέπει να τους αξιοποιούμε στο έπακρο. Ο προϋπολογισμός μας ε, είναι αρκετά περιορισμένος ε, για τα θέματα αυτά. Οπότε δεν μπορούμε πάντα να εγγυηθούμε τη δυνατότητα μετάφρασης όλων των εγγράφων της Europol σε όλες τις γλώσσες σύμφωνα με το γλωσσικό μας καθεστώς όλα τα έγγραφα που κατατίθενται ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι γραμμένα στα αγγλικά. Όλα τα νομικά έγγραφα και οι αποφάσεις μας δημοσιεύονται επίσης στα αγγλικά. Εκτός αν πρέπει να ε, δημοσιευθούν και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί ε, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα. Συμπεράσματα. Τι σχεδιάζουμε για το μέλλον. Στις 3 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση. Τα θέματα προς είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων, ενδεχόμενες εξελίξεις ε, στο θέμα αυτό, συνεργασία με τους εταίρους προτεραιότητας, η συνεργασία μας με την Ιαπωνία, με το κέντρο το παρατήρηση των ναρκωτικών και άλλα σημαντικά θέματα και άλλους σημαντικούς οργανισμούς. Επίσης, θα αποφασίσουμε ποιος θα είναι επόμενος πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Και σε ό,τι αφορά ε, επίσης το προσωπικό, ε, τον κανονισμό, το δημοσιονομικό, μάλλον το, υπηρεσιακής κατάστασης, ε, για τη μεγαλύτερη διαφάνεια, για το πόθεν έσχεστο στο μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Όλα αυτά σύμφωνα με τους ε, κανόνες που ισχύουν και την κειμένη νομοθεσία. Και όπως είπε και ο κύριος Βάιντιγκερ από την ε, Αυστρία, στις 4 Οκτωβρίου τα διοικητικά συμβούλια Ευρωπόλ και Frontex θα έχουν κοινή συνεδρίαση για να συζητήσουν τα περαιτέρω βήματα μιας πιο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και οι δύο οργανισμοί αυτοί έχουν συμπληρωματικές εντολές και η Ευρωπόλ και ο Frontex έχουν να διαδραματίσουν ε, αυξημένο ρόλο στο μέλλον για την ε, συντονισμένη απάντηση στη διακίνηση ανθρώπων και στη διακίνηση μεταναστών. Θα συζητήσουμε επίσης και για τη μελλοντική μας διαλειτουργικότητα, δηλαδή των συστημάτων πληροφοριών που έχουμε. Και οι δύο οργανισμοί σίγουρα δεν μπορούν παρά να ενισχυθούν με, τη συνεργασία. Κατά την άποψή μου, ε, αυτές ε, οι εξελίξεις θα έχουν ένα καταλητικό ρόλο για τη λειτουργία της Ευρωπόλ. Στο μέλλον θα μπορούμε να υποστηρίζουμε το Frontex, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και επίσης η Ευρωπόλ θα έχει ευρύτερη πρόσβαση σε ε, αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα είναι πιο αποτελεσματική στον υποστηρικτικό ρόλο που διαδραματίζει προς τις διοκτικές αρχές των κρατών μελών. Θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να ε, βοηθούμε στη συνεργασία με σκοπό την πρόληψη και την επάταξη του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος στην Ένωση και της τρομοκρατίας. Αυτά! Και σταματώ εδώ με χαρά ε, να σας ενημερώνω και στο μέλλον ε, για τις δραστηριότητε μας και με χαρά θα ακούσω και τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσω σε αυτές. Είπα στην αρχή ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Γι' αυτό ε, μίλησα χωρίς να κάνω καμία εισαγωγή. Προσπαθώ να τα πω με μεγάλη συντομία. Ευχαριστώ που με καλέσατε, πάση περιπτώσει, γιατί δεν το είπα στην αρχή για λόγους χρονικούς. Η Πρόεδρος, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πάρκνα, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί στη σύνοψή σας αναφερθήκατε και στα προβλήματα ε, που υπάρχουν τώρα αυτές τις παιδικές αρρώστιες της συνεργασίας που είναι στα Σπάργανα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τσβετάνοφ ε, για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του για τα πεπραγμένα ε, της τελευταίας περίοδου. Παρακαλώ. Ε, αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σημειώσω ότι με χαρά συμμετείχα στην 107η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ ως συμπρόεδρος της ΜΟΚΕ. Πριν πω στα συγκεκριμένα σημεία που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ε, της παρουσίας μου εκεί, θα ήθελα να σας πω ότι ως εκπρόσωπο της ΜΟΚΕ ε, δέχθηκα μεγάλη και εγκάρδια υποδοχή από όλους τους ειρανωτές και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διευθύντρια και σας ευχαριστώ για αυτό. Ε, ο κύριος ε, Πάρκνα ε, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό που απίφθηνα σε αυτή τη συνεδρίαση. Θεωρήθηκε ανοιχτό και ειλικρινή και η κυρία Ντεμπόλ μίλησε για τον κανονισμό της Ευρωπόλ που δίνει σημαντικό ρόλο στου βουλευτές και το θεωρεί αυτό σημαντικό για να βελτιωθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια ε, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επίσης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπόλ να διατηρεί την επαφή της μαζί μας και δεσμεύτηκε ότι θα συμμετέχει στις εργασίες μας. Εγώ όπως σας είπα συμμετείχα στις 4 Μαΐου σε αυτή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρθηκα μόνο ε, σε ένα σημείο που έχει να κάνει με τη συμμετοχή της ΜΟΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας αυτής, της μικτής, είναι ακριβώς η λογοδοσία και η ε, νομιμοποίηση της Ευρωπόλ στην καθημερινή δουλειά και στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό τόνισα ότι αυτά που αναφέρουν ε, το, η αιτιολογική σκέψη 20 και ε, το άρθρο 14 παράγραφος 4 του κανονισμού της Ευρωπόλ σχετικά με την παρουσία μέλους της ΜΟΚΕ θα πρέπει να ερμηνεύονται με την ευρία έννοια, την ευρύτατη δυνατή και αυτό πιστεύουν το, και οι άλλοι συμπρόεδροι. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού μας, ε, καλούμε θα ως παρατηρητές ε, ε, χωρίς δικαίωμα ψήφου τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω αυτό να αφορά και όλες τις μελλοντικές συνεδριάσεις. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο μίλησα, είπα ότι οι συμπρόεδροι περιμέναμε να ε, αναφέρεται και να αντανακλάτε το άρθρο 51 του κανονισμού της Ευρωπόλ. Βεβαίως τηρουμένου πάντα όλων των διατάξεων για την εχεμήθεια και το απόρριτο. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων οι συμπρόεδροι της ΜΟΚΕ και ε, ο πρόεδρος ε, του εκτελεστικού του Διοικητικού Συμβουλίου μάλλον για να δούμε με ποιο τρόπο ο εκπρόσωπος της ΜΟΚΕ θα ενταχθεί σε αυτό το σχήμα και θα συμμετέχει. Επίσης, πρότεινα μέχρι να οριστεί επίσημος εκπρόσωπος ΜΟΚΕ να υπάρξει συνέχεια της τρέχουσας πρακτικής. Δηλαδή, να απευθύνεται πρόσκληση στους συμπροέδρους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άλλα θέματα που ανέφερα στην παρέμβασή μου ήταν ε, να επανεξετάσουμε το θέμα το γλωσσικό δεν μπορεί να είναι μόνο στα αγγλικά τα κείμενα. Αγγλικά και γαλλικά είναι επίσημες γλώσσες της ΜΟΚΕ και ελπίζω ε, στο μέλλον το, το Διοικητικό Συμβουλίο να μας απευθύνει την αλληλογραφία σε αυτές τις δύο γλώσσες τουλάχιστον. Επίσης αναφέρθηκα και στο χρονοδιάγραμμα και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα εργασιών για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισμού Ευρωπόλ. Υπό την έννοια αυτή, κάλεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ να προτείνει ένα κοινό χρονοδιάγραμμα εργασιών για τη διαβούλευση σχετικά με το πολιετές πρόγραμμα. Για τα θέματα τώρα της εχεμήθειας ή της εμπιστευτικότητας, του ζήτησα να συμφωνήσουν με τη γραμματεία της ΜΟΚΕ για να δούμε ποιο είναι το καθεστώς κάποιων εγγράφων ε, που δίνει στις συνεδριάσεις ε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, τόνισα ότι οι συνεδριάσεις της ΜΟΚΕ αποτελούν καταπληκτική ευκαιρία για θεματικές συζητήσεις σε πολλά ε, θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν με ε, τις εργασίες της Ευρωπόλ και τους εξωτερικούς εταίρους και την εξωτερική ε, στρατηγική. Στην τελευταία λοιπόν συνεδρίαση στη Σόφια το Μάρτιο της μεικτής ομάδας ήμασταν εμείς οι διοργανωτές και είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε σχετικά με τις ε, πρόσφατες εξελίξεις στη συνεργασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και τα σχέδια για την ενεργή ένταξη των χωρών αυτών στην αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συζήτηση υπήρξε αντίδραση στη δική μου παρέμβαση και το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο της εχεμήθειας και της εμπιστευτικότητας και μα ζήτησε να έχουμε κατανόηση γιατί ορισμένα έγγραφα δεν δημοσιεύονται, Αλλιώ απειλούν ε, τρέχουσες επιχειρήσεις. Επίσης σημείωσα ότι το άρθρο 14 του κανονισμού δίνει ε, αρκετή ευχέρεια κινήσεων ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους προσκεκλημένους παρατηρητές. Ο κύριος Πάρκνα τόνισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα παίρνει, να παίρνει αποφάσεις από κοινού και κάλεσε τους εθνικούς εκπροσώπους να τα συζητήσουν αυτά τα θέματα με τις υπηρεσίες τους και τα κοινοβούλια τους για να αρχίσει αμέσω η νέα διαδικασία έτσι ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να συζητηθεί το θέμα με τα λόγου γνώσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποκρισταλώσει ε, θέση σχετικά στη συνεδρίαση του του Οκτωβρίου και ε, θα μας ε, στείλει μια επιστολή για να μας ενημερώσει. Εγώ επίσης τόνισα ε, ως παρατηρητής στη συνεδρίαση αυτή ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπόλ και για όλους τους βουλευτές να διατηρηθεί η απρόσκοπτη συνεργασία μας. Είμαστε μια μεικτή ομάδα που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αποτελέσουμε εμπόδιο ε, για τον οργανισμό. Ίσα ίσα θέλουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική την Ευρωπόλ με ένα διάλογο επικοδομητικό, γόνιμο, χωρίς εμπόδια και προσκόμματα. Ελπίζω να συνεισέφερα από πλευρά μου στο διάλογο αυτό μέσω τη συμμετοχή μου στη συνεδρία τη 4 η Μαΐου και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και την κυρία Ντεβόλ για το επικοδομητικό πνεύμα καθώ επίση και του συναδέλφου, ε, βουλευτέ από όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσβετάνοφ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή, την παρουσίασή σας τι μας δείχνει αυτό. Πόσο αγαστή είναι η συνεργασία μας με όλα τα θέματα που μπορεί ίσως στο μέλλον να διαμορφωθούν καλύτερα. Αλλά είμαστε ένα τόσο νέο όργανο που πραγματικά πρέπει να περάσουμε αυτές τις παιδικές ασθένειες και την άλλη φορά να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ε, ακολουθεί η συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο. Από την Κύπρο. Ο κύριος Μυριάνθους, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσβεστάνοφ για τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟΚΕ που μετέφερε κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαΐου. Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω ότι η εκλογή ενό αντιπροσώπου τη ΜΟΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπω προβλέπει ο κανονισμό λειτουργία μα, θα ενίσχυε το θεσμό διασφαλίζοντα την αναγκαία συνέχεια τη παρακολούθηση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίση, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τι δραστηριότητε του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τι συνεργασίε με την Αιγυπτών καθώς και με άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής από τις οποίες παρατηρούνται εισδροές μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο. Παρακαλώ τους ε, δύο ομιλητές μας. Εσείς πάλι να απαντήσετε κύριε Πάρκνα. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως ήδη είπα και στην ομιλία μου, για το Διοικητικό Συμβούλιο, η συνεργασία με την ομάδα σας, την ΜΟΚΕ, την Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, είναι πολύ σημαντική. Και ήδη βλέπουμε τα θετικά της συνεργασίας αυτή, τα ωφέλη. Δυστυχώς όμως σήμερα σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω. Δεν μπορώ να προδικάσω την τελική απόφαση που θα ληφθεί. Αυτό, αυτή η συζήτηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα σα ενημερώσω στο δυνατόν συντομότερα. Ε, ότι σε ό,τι αφορά τι διαφορετικέ επιχειρησιακέ δράσει τη Ευρωπόλη, Η εκτελεστική διευθύντρια σας έδωσε ήδη μια διεξοδικότατη επισκόπηση και για το πρόγραμμα συνεργασίας με την Τουρκία και γενικότερα για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Βεβαίως για την Ευρωπόλη και το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι άκρο σημαντικό να έχουμε αγαστές σχέσεις και για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τις επιχειρησιακές μας ε, δράσεις. Είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα την τρομοκρατία χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίε. Ο καθένα το καταλαβαίνει αυτό. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπόλ. Όμω πρέπει να είμαστε και πιστοί να τηρούμε το νομικό πλαίσιο, τους κανόνες. Ε, δυστυχώς δεν το έχουμε ε, σχεδιάσει εμείς όπως μας βολεύει το πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσφετάνοφ, θέλετε να πείτε τίποτα έτσι, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη Εμένα μου είχε ζητηθεί να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, να σας αναφέρω ότι έγινε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τηρώ αυτό και σταματώ στη συμφωνία που είχαμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρίσω το πέρα της συζήτηση αυτής. Έχω να σας ανακοινώσω ότι ε, ολοκληρώνουμε την πρώτη ημέρα ε, της ε, συνεδρίασής μας και σας προσκαλώ στη δεξίωση που θα παρατηθεί στον χώρο Γεχούντι Μενουχίν που είναι ακριβώς από κάτω στο δεύτερο όροφο και έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε βιενέζικο κρασί παρακαλώ ε, συνεχίζοντας τις συζητήσεις. Είστε προσκεκλημένοι, ε, έχετε ε, στη θέση σας και πασατέμπο που έχουμε από τη Στηρία ε, και μπορείτε να απολαύσετε τα προϊόντα της Αυστριακής Προεδρίας. Ε, αύριο θα με αντικαταστήσει ο συνάδελφος Μπούχμαν και θα συμπροεδρεύσει διότι εγώ δυστυχώς αύριο πρέπει να επιστρέψω στη Βιέννη πρωί-πρωί και η αυριανή σας λοιπόν συνεδρία αρχίζει στις 9.30 ώρα στην απέναντι αίθουσα PHS 3C50, όχι εδώ στο ημικύκλιο, ακριβώς απέναντι ε, την αίθουσα της Ολομέλειας. Ε, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, καλό μας βράδυ. Και καλή επιτυχία και συνέχεια ε, στην αυριανή ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.